I think Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που είστε τόσο πολύ για την τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις διακοπές. Βελτίωση των συνδέσεων και της πρόσβασης στις ε, υποδομές μεταφορών στην ε, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έκθεση πρωτοβουλία, εισηγητή ο Τόμα Πιότρε Πόρτσιεβα, στον οποίο και το λόγο. Κυρίε και κύριοι, δεύτερη φορά συζητάμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας και αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης στις υποδομές μεταφορών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ιδίως από την Επιτροπή Μεταφορών. Όσους λοιπόν ε, υπέβαλαν τροπολογίες, αλλά και προτάσεις γενικά και εμπλούτησαν την έκθεσή μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Με βοήθησαν πάρα πολύ. Η έκθεσή μου έτσι έγινε ένα στρατηγικό κείμενο. για να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις η κεντρική και η ανατολική Ευρώπη σε θέματα μεταφορών. Οι προκλήσεις αυτές είναι όντως αντιμετωπίσιμες. Χάρη και στις συστάσεις που κάνατε και τις οποίες περιέλαβα στην έκθεσή μου. Σήμερα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους συντονιστές των ε, ομάδων για να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα τα ξαναπούμε με τους συντονιστές και χαίρομαι ιδιαίτερους που γενικά υπάρχει πολύ καλή και επικοδομητική διάθεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων για να καταλήξουμε σε συνενετικές διατυπώσεις για τις κατευθύνσεις ανάπτυξης των μεταφορών, τους ε, στρατηγικούς στόχους που πρέπει να υλοποιήσουμε. Οπότε σήμερα δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαμε και στην προηγούμενη συνάντηση, όταν σας παρουσίασα για πρώτη φορά την έκθεσή μου, θα προτιμούσα να ακούσω τις δικές σας παρατηρήσεις, να ασχοληθούμε κυρίως με τις παρατηρήσεις και τροπολογίες σας. ούτως ώστε να μπορέσω να τις ε, συμπεριλάβω ακόμη καλύτερα στο κείμενό μου. Γι' αυτό είμαι στη διάθεσή σας και σας παρακαλώ να μου κάνετε περτέρω παρατηρήσεις και θα κάνω ό,τι μπορώ ούτως ώστε να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ για να γίνει στρατηγικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο πρόεδρο. Τώρα, Άντορ Ντέλη. Ευχαριστώ. Το σχέδιο ήταν ήδη μια πάρα πολύ καλή αφετηρία και βελτιώθηκε με τις ε, τροπολογίες των συναδέλφων. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω την πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Πορέβα και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές, γιατί είναι σαφές ε, ότι είχαμε ήδη σήμερα μια πάρα πολύ καλή συνάντηση και καλύψαμε σχεδόν τους μισούς από τους 34 ε, συμβιβασμούς. Αναμένω και την επόμενη συνεδρίαση μετά τις διακοπές και ελπίζω να μπορέσουμε να τηρήσουμε την προθεσμία που είχε τέθει 26 Σεπτεμβρίου δηλαδή για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Είναι προφανές ε, πως οι υποδομές ε, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί μετά από μια δεκαετία και πάνω ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στις χώρες μας. Συμφωνούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη πηγαίνει χέρι-χέρι με τις καλές υποδομές, οπότε θα πρέπει βεβαίως οι επενδύσεις να κατευθυνθούν κυρίως σε αυτές τις χώρες. Αλλά οι επενδύσεις αυτές θα ωφελήσουν και άλλες χώρες και οικονομίε οικονομίες και οι διάδρομοι διευρωπαϊκών δικτύων παίζουν ένα κρίσιμο ρόλο εδώ πέρα. Και δεν μπορούμε να έχουμε ένα φαινόμενο διαδρόμου χωρίς να γίνουν οι επενδύσεις στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον πρέπει να εστιάσουμε στο συνολικό δίκτυο για να αποφύγουμε τις στενοπούς Επιπλέον, η έκθεση σωστά τονίζει τον ρόλο περιφερειακών έργων όπως η Καρπαθία ή η Βαλτική Οδός και επίσης οι διασυνδέσεις με την Ανατολική Γειτονία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Έχοντας κατά νου τις τεράστιες οικονομικές ανάγκες, είναι σαφές πως τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να βρουν όλα αυτά τα λεφτά μόνα τους. Και υπάρχουν καλά στοιχεία στην έκθεση για την χρηματοδότηση που ενισχύονται περαιτέρω με τις ε, τροπολογίες ειδικά όσον αφορά την χρήση του στρατηγικού ταμείου και του μέσου συνδέοντας στην Ευρώπη και η ανάμειξη της χρηματοδότησης επίσης αναφέρεται. Οπότε αναμένω την συνεργασία με τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις ε, εισηγητές και ελπίζω να έχουμε καλές διακοπές γιατί ήδη πηγαίνουμε αρκετά καλά. Ευχαριστώ. Κλαόδιο Ταπαντέλ. Κλαουδία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για το σχέδιο έκθεσης, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πορέμπα. Να ευχαριστήσω βέβαια και τους υπόλοιπους εισηγητές, τους σκιώδες εισηγητές για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε ένα στρατηγικό κείμενο το οποίο θα καταφέρει να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ασχοληθεί λίγο περισσότερο με τον εξυγχρονισμό των μεταφορικών υποδομών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τις τροπολογίες, οι υποδομίες και οι υποδομές με και η διασυνδεσιμότητα στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ σημαντική για τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφορικές υποδομές αντιστοιχούν στον ίδιο τον πυρήνα της οικονομικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποτελεσματικές μεταφορικές υποδομές. Οι συνάδελφοι από τις πολιτικές ομάδες υπέβαλαν τροπολογίες και η δική μου πολιτική ομάδα βέβαια. Θα ήθελα να τονίσω την εξή όμω ιδέα. Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξη, λαμβάνοντα υπόψη όλε τι πτυχέ που έχουν να κάνουν με τι υποδομέ μεταφορών. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να αφορά όλου του τρόπου μεταφορών και θα πρέπει να στοχεύει και στη δημιουργία βιώσιμων διασυνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει και ένα ακόμα σημείο το οποίο πρέπει να θίξουμε, το σχέδιο RTET e της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, TEN-T, και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε καταρχάς κάνοντας επενδύσεις σε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση του δικτύου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα το δίκτυο των Δυτικών Βαλκανίων, και αυτό αναφέρεται και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αναφέρονται στην ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη. Συμφωνούμε ότι όντως εδώ πέρα πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο την εσωτερική ναυσιπλοεία, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Όσον αφορά τώρα τους στόχους για τις υποδομές αυτές καθ' αυτές, Έχουμε υποβάλει και εμείς και άλλες πολιτικές ομάδες κάποιες τροπολογίες που αναφέρονται στα χρηματοδοτικά μέσα με τις πολλές διαφορετικές μορφές επιδοτήσεων που μπορεί να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαιρετίζουμε το ότι αυξάνεται ο αριθμό των χρηματοδοτικών μέσων και ότι εμπλέκεται όλο και περισσότερο ο ιδιωτικό τομέα. Θα θέλαμε να τον βοηθήσει βέβαια τον ιδιωτικό τομέα και η ίδια η διοίκηση των κρατών μελών. Ορισμένα κράτη-μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης χρειάζονται και τεχνική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να καταφέρουν να υλοποιήσουν συγκεκριμένα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια. Από την άλλη, ορισμένοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο υψηλό ποιοτικό επίπεδο των υπηρεσιών μεταφορών, ότι το, η ποιότητα πρέπει να είναι πολύ ψηλή προς το συμφέρον των καταναλωτών και αναφέρεται επίση και ο τουριστικό κλάδο. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που σχετικά με τον κλάδο αυτό υπευλήθησαν τροπολογίε και από την πολιτική μου ομάδα και από άλλε πολιτικέ ομάδε. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι έχει συμπεριλάβει ο συγητή αυτέ τι τροπολογίε στι συμβαστικέ του προτάσει. Πρέπει να αναγνωριστεί η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών. Μετά τη δεύτερη διαπραγμάτευση που θα, εξαχθεί, Είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε να συντονίσουμε περισσότερο την προσέγγισή μας και θα καταλήξουμε κατά αυτόν τον τρόπο σε μια κοινή τοποθέτηση ιδιαίτερα θετική και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιάννος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξ ονόματος του κυρίου Τελίτσκα την να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία και την εξαιρετική αυτή έκθεση και τις ε, καλές συμβιβαστικές προτάσεις. Όλοι οι βουλευτές από όλες τις ομάδες κατέθεσαν διάφορες ε, τροπολογίες ε, που θεωρούμε ότι βελτιώνουν το κείμενο. Θα ήθελα να φέρω και εγώ κάποιες και να ζητήσω στήριξη των συναδέλφων. Στην παράγραφο 9 Θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να εξετάζει και να κοιτάει, αλλά να λάβει υπόψη το πώς θα μπορούν να διαμορφωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στα Βαλκανικές χώρες Ανατολικής Γειτονίας στην Ουκρανία. Μετά στο άρθρο 11α θέλουμε να υπάρξει ψηφιοποίηση της υποδομής των μεταφορών και έχουμε καταθέσει μια τροπολογία στο άρθρο 17 όπου ζητάμε από τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν το σύστημα ERTMS ε, για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Γιατί έτσι θα υπάρχουν λιγότερα προβλήματα στις συνοριακές ε, διαβάσεις. Μετά τροπολογία στο άρθρο 21 έχουμε που μιλάμε για την συμφωνία που υπάρχει για τον Δούναβη από το 1946 είναι πλέον ξεπερασμένη και έτσι περιορίζει την πλοημότητα του Δούναβη και θα δούμε το τι μπορεί να γίνει για να ξεπεραστεί αυτή, για να επανεξεταστεί αυτή η ξεπερασμένη συμφωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι και τον Σεπτέμβριο. και να έχουμε μια σωστή έκθεση στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, θα μιλήσω και εγώ, θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπατε, την πλοημότητα του Δούναβη, έχουμε την συνθήκη του 1946 που πρέπει να επανεξεταστεί, αλλά και πριν από... και πριν από 30 χρόνια ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και αυτό πρέπει να λάβω Εγώ είχα πάει με ένα κανό από το Ίγκροστάτ στη Μαύρη Θάλασσα και πρέπει να προσέχει κανείς με το κανόμι τον παρασύρουν τα κύματα και τα, τα απόνερα. Όταν περνάει μεγάλο καράβι. Πριν από τρία χρόνια πάλι το ίδιο έκανα 100 χιλιόμετρα στον Δουναβί, είδα τρία πλοία. Το Σαββατοκύριακο στην Πρατισλάβα έφαγα ε, στις όχθες του ποταμού δεν είδα κανένα πλοίο, μόνο πλοία που έκανε κουραζιέρες και επιβατικά. Τα κανονικά πλοία λοιπόν μπορούν να περάσουν, μόνο τα τεράστια δεν χωράνε. Γιατί είχαμε φτιάξει τότε στη Γερμανία, είχαμε σκεφτεί τότε στη Γερμανία ένα κανάλι Rhein-Main-Dunavi, αλλά μας είπε ο, μεγαλύτερο, ο, είπε ο Υπουργός ε, ε, Συγκοινωνιών ότι ήταν μεγαλύτερη βλακή από τον πύργο της Βαβέλ. Γιατί, γιατί δεν υπήρχαν πλοία. Αλλά θα ήταν τεράστια επιτυχία αν είχαμε προβλέψει το 10% της ε, κίνησης της σημερινής. Πρέπει λοιπόν να λάβουν υπόψη ότι στην εσωτερική ναυσιπλοεία τα τελευταία 20 χρόνια μειώθηκε αυτή από το 20% στο 8% και το 80% έχει περιοριστεί στον Ρήνο. Οπότε να επεκτείνουμε τον Δούναβη προς βορρά έχει ξεπεραστεί πλέον και η Βαβαρία που το ζήταγε το έχει ξεχάσει, στην Αυστρία υπήρχαν διαδηλώσεις. Δεν χρειάζεται και, και δεν πρόκειται να προχωρήσει κιόλας. Αλλά μπορώ να σας πω γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Στη Γερμανία έχουμε ανα πλοίο της εσωτερικής ναυσιπλοείας τρία άτομα στην διοίκηση. Οπότε πρέπει να δικαιολογήσουν την ύπαρξή του και βγάζουν συνεχώ νέου κανόνε. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού θα επενδύσουμε. Είμαι υπέρ τη εσωτερική ναυσιπλοεία, αλλά πρέπει τα πλοία να προσαρμοστούν στον ποταμό και όχι αντιστρόφω. Και πρέπει να επενδύσουμε εκεί όπου υπάρχει όφελο μετά τι αρνητικέ εμπειρίε που είχαμε. Δεύτερον, εκεί όπου μπορούν να γίνουν τα πράγματα με λίγα λεφτά ή με καθόλου λεφτά, ε, δεν είναι τόσο στα βαλκανικά κράτη, αλλά στη σύνδεση με αυτό την πρώην Δυτική Ευρώπη. Σας είπα πριν για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Βρατισλάβας για τα τέσσερα ε, χιλιόμετρα. Από το Βαλκύρχεν στο Νόβο Ούντελι μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας επίσης 25 χρόνια δεν έχει υπάρξει μια ανακαίνιση της διαδρομής που είχε καταστραφεί επί παραπετάσματος. Λοιπόν, δεν πρέπει να συνδέσουμε μόνο τα Βαλκάνια εσωτερικά, αλλά και με την Δυτική Ευρώπη να αποκατασταθούν οι συνδέσεις. Εκεί πέρα δεν χρειάζονται πολλά λεφτά. Αυτό το οποίο λείπει είναι πολιτική βούληση. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Βιμ Φαντεκάμπ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Με την ε, κύρια Ντελή ήμασταν ε, στις, ε, στο Ρότερνταμ στις 10 Days και μιλήσαμε για την βυθοκόρηση, για το εάν είναι κάποια συντήρηση ή επένδυση. Και βρισκόμαστε τώρα σε μια φάση των συμβιβαστικών προτάσεων, αλλά θα ήθελα να πω, να ρωτήσω την Κομισιόν, εάν η βυθοκόρηση του Δούναβη θεωρείται επένδυση ή απλώς συντήρηση. Γιατί πολλά κομμάτια, σε πολλά κομμάτια έχει επικαθίσει η άμμος. Λοιπόν, μετά έχουμε την τροπολογία 46 της κυρίας Γραπίνη. Εκεί πέρα λέμε πως τα περισσότερα έργα του ΕΦΣΙ είναι στη Δυτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς γίνεται αυτό. Βλέπω σε άλλες ε, τροπολογίες που ζητάμε περισσότερη έμφαση στο ταμείο αυτό και εξακολουθεί βεβαίως στην Ανατολική Ευρώπη να δίνεται βάρος στις επιχορηγήσεις και λιγότερο στα δάνεια, στα δάνεια του ΕΦΣΗ. Ίσως αυτό το στοιχείο θα μπορούσε να ενισχυθεί στο συμβαστικό κείμενο. Αυτά ευχαριστώ. Danke sehr. Olga Selanova hat sich nochmal gemeldet. Όλγα Σελάνοβα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σίτη. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση, ήμουν Και έχω συντάξει και τη λευκή βιβλίο για τις μεταφορές. Και έχει υποθεί ότι πρέπει να υπάρξουν ισότιμες συνθήκες ε, μεταξύ των παλιών και των νέων κρατών. Χαίρομαι που αυτή η διατύπωση συμπεριλαμβάνεται και στην παρούσα έκθεση. Υπέβαλα μια σειρά από τροπολογίες και θα μπορούσα ίσως να τονίσω ότι η βελτίωση της ε, πλοηγησιμότητας των εσωτερικών υδατίνων οδών δεν αφορά μόνο το, το Δούναβι αλλά και τον Έλβα. Θα ήταν καλό να βελτιώσουμε την κατάσταση συνολικότερα. Και θα ήταν σκόπιμο να πάμε στην Τσεχία το Σεπτέμβριο για να δούμε επιτόπου την κατάσταση. Χρειαζόμαστε υψηλή ε, ποιότητας υποδομές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς σιδηροδρόμους. Υπάρχει μεγάλο κενό δεν έχουμε αρκετές γραμμές υψηλής ταχύτητας. Και κάτι άλλο που θέλω να θίξω, που περιλαμβάνεται στην έκθεση, αλλά θα ήθελα να τονιστεί περισσότερο, είναι ο συντονισμός και συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στη φάση προπαρασκευής και προγραμματισμού διαμεθοριακών συνδέσεων, ούτως ώστε να έχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους και να δώσουν πραγματικά ωφέλη. Και πάλι ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Harold Kreuters. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζουμε την έκθεση και την εργασία που έκανε ο συγητής και η Σκιώδης και αυτά που αναφέρουν για τις ανάγκες ε, της περιοχής αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Επίσης, ε, η σημασία της διαλειτουργικότητας και του ATMS είναι καλοδεχούμενα όλα αυτά. Η έκθεση αυτή θα ήθελα να κάνω έκκληση να μην ε, εστιάσει υπερβολικά συγκεκριμένα προγράμματα. Τα ten μας δίνουν ένα συνολικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας υποδομής στην Ευρώπη που μέχρι το, ε, το 2030 θα ε, μας δώσει ένα πλήρως λειτουργικό δίκτυο. Για την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη υπάρχει πολύ καλή απορρόφηση από τα κράτη-μέλη. Ήδη έξι κράτη-μέλη έχουν αξιοποιήσει 100% τις συνολικές τους χρηματοδοτήσεις και θα υπάρξει άλλο 1,1 δις που θα, που θα προκηρυχθεί ε, το φθινόπωρο και θα επανέλθω στην Επιτροπή σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Από τον Οκτώβριο λοιπόν το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτήσεων για τις χώρες αυτές θα προκηρυχθεί. Πολύ καλή απορρόφηση λοιπόν και σίγουρα τα 11,3 δις θα δαπανηθούν πλήρως μέχρι τέλος του χρόνου ή τουλάχιστον θα δεσμευθούν πλήρως. Επίσης πρέπει να δουν και τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του ΕΦΣΥ. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και το ΕΦΣΥ. Και θα απευθυνθεί 15 χώρες συνοχής. Στο φθινόπωρο θα τις επισκεφθούμε μία-μία για να τις βοηθήσουμε να αξιοποιήσουν και προϊόντα του ΕΦΣΥ. Νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει για ορισμένα προγράμματα. Προγράμματα πυρήνα ή προγράμματα, ε, συγγνώμη, προγράμματα λιμένων ή προγράμματα αυτοκινητοδρόμων. Επίσης χρειαζόμαστε σταθερότητα δεν θέλουμε να αναφέρουμε πολλά προγράμματα. Ήδη είναι αρκετά μακροσκελή η κατάλογη. Χρειαζόμαστε δύο περιόδου πολιτών προπτικών για να εκτελεστούν αυτά τα προγράμματα και χρειάζεται συνέχεια μεταξύ του 2014 και του 27. Γιατί πολύ συχνά μα έχουν επικρίνει ότι αλλάζουν συνεχώ οι προτεραιότητε και κανένα επενδυτή δεν μπορεί να παρακολουθήσει κάτι τέτοιο τόσο ώστε να μα βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν επίσης διάδρομοι το είπε και η κυρία Σεναλόβα για τον συντονισμό και τη συνεργασία. Έχουμε διαδρόμους που διασχίζουν Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο την περιοχή. Άρα πρέπει να μα στηρίξετε ως Επιτροπή για να εφαρμόσουμε τους διαδρόμου Και χαίρομαι που πάντα αντιμετωπίζετε τόσο σωστά αυτό το θέμα. Οι συντονιστέ παρουσίασαν και στο Ρότερνταμ το πρόγραμμα εργασιών και θα ήθελα παρακαλώ να μελετήσει η Επιτροπή σας και το δεύτερο ε, πρόγραμμα δράσης και εκεί θα διαπιστώσετε ότι οι προτεραιότητες που έχετε αποφασίσει μαζί με τα κράτη-μέλη τώρα εφαρμόζονται. Επίσης, να σα ενημερώσω και τον κύριο Φαντεκάμπ και τον εισηγητή. Η βυθοκόρηση ορισμένες φορές μπορεί να συγχρηματοδοτηθεί από εμά, όχι η συνήθι συντήρηση, αλλά η δημιουργία των ε, προποθέσεων για τη βυθοκόρηση βεβαίω μπορεί να χρηματοδοτηθεί και από εμά. Αυτό θα βοηθήσει ε, την πρόοδο στο Δούναβι. Και έχετε δίκιο. Δεν χρειάζεται παντού να έχουμε ε, τις ε, απόλυτες δυνατότητες. Μπορούμε να βρούμε νομίζω καλές λύσεις και για το Δούναβι. Ούτω ώστε να υπάρχει πλογισμότητα. Αυτά πρόεδρε. Και βεβαίω με χαρά θα παρακολουθήσουμε και την περαιτέρω συζήτηση, ούτω ώστε να αξιοποιήσουμε την έκθεση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, και ο Πρόεδρο. Και τώρα ο Τόμας Ποτσέμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους. Τα όσα αναφέρετε πραγματικά θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για μένα στην μελλοντική μου εργασία και θα τα λάβω πλήρως υπόψη μου κατά την προετοιμασία των συμβαστικών προτάσεων. Να πω και κάτι ακόμα όμως. Η έκθεση αυτή έχει πολλούς διαφορετικούς στόχους, ένας εκ των οποίων είναι να ενισχύσει και να τονίσει τη σημασία της δημιουργίας μεταφορικών υποδομών στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Και θα πρέπει να μείνουμε εδώ στο ζήτημα της ασφάλειας για τις υποδομές αυτές. Το είχα τονίσει αυτό και σε συζητήσεις που είχα με σας είναι σημαντικό να στείλουμε και το μήνυμα αυτό. Μια καλύτερα διαστεδεμένη Ευρώπη είναι και μια πιο ασφαλής Ευρώπη. Να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πληροφορίες που μόλις τώρα μας έδωσε. Θα έρθω άμεσα σε επαφή μαζί σας, σε προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να καταφέρουμε να ανταλλάξουμε περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες θα μπορέσω συνέχεια να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου. Υπάρχει ένα σημείο όμως με το οποίο διαφωνώ. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα λεπτομερής η έκθεση αυτή, ότι δεν θα πρέπει να επιστέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Στόχος της έκθεσης είναι να προβάλλει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα των μεταφορών. Προσπάθησα λοιπόν να αφαιρθώ σε συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένους στόχους που εμείς ως ευρωβουλευτές θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο ή λεπτομερή προβλήματα τα οποία θα μπορέσουμε εμείς να αντιμετωπίσουμε, περιοχές δηλαδή στις οποίες δεν υπάρχουν απαραίτητες υποδομές. Για άλλη μια φορά πάντως θα ήθελα να σε ευχαριστήσω τον, όλους τους και οδησηγητές και όλους τους συναδέλφους και τον πρόεδρό μας βέβαια για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και το Σεπτέμβριο όταν θα σας δω πάλι εκ νέου. Θα έχουμε ξεκουραστεί τότε και θα είμαστε σε θέση πια να εκπονήσουμε μια έκθεση η οποία θα είναι μια πραγματική στρατηγική έκθεση για την πολιτική μεταφορικών υποδομών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Η προθεσμία για την ψηφοφορία, μάλλον η ημερομηνία της ψηφοφορίας είναι 26 ε, Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε διακοπή τώρα, γιατί θα έχουμε κάποιους ομιλητές. Θα συνεχίσουμε στις 4 λοιπόν. Πρέπει να σας πω όμως ότι ο Κρίστοφα Φόρντ από τη γραμματεία της Τραν μας αφήνει. Εργάστηκε μαζί μας εδώ και 7 χρόνια και πρέπει να πω ότι ήταν θαυμάσια συνεργασία και πολύ ευχάριστη και λυπάμαι ιδιαίτερα. Απλώς ε, πρέπει να τον αφήσουμε για να μας φύγει, να μας πάει στην Επιτροπή Έμπλα. Οπωσδήποτε θα βοηθήσει την Έμπλα, αλλά εμείς θα, εμάς θα μας λείψει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε και του εύχομαι κάθε επιτυχία στην Επιτροπή Απασχόλησης και σίγουρα θα βοηθήσει και εκεί όπως και εδώ. Και νομίζω ότι από πλευράς όλων που συνεργάστηκαν μαζί του μπορώ να του, ζητήσω, να του πω ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Und jetzt machen wir eine kleine... Λοιπόν, μία μικρή διακοπή για να μπορέσει να πει το καφέ το ΒΙΜ και θα συνεχίσουμε στις 4.

Ja, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, σα καλωσορίζω θερμά στη συνέχιση της συνεδρίασή μας. Την τελευταία πριν από τις διακοπές Περνάμε τώρα στην ειδική ομάδα τουρισμού ανταλλαγή απόψεων για τη χρήση ενωσιακών πιστώσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στον τουρισμό. Πριν αρχίσω τη συζήτηση, να πω ευθύ εξ αρχή ότι το θέμα τη συνεδρίασή μα σήμερα είναι ιδιαίτερα σκόπιμο. Υπάρχει ένα θέμα που τίθεται σε όλες μας τις συνεδριάσεις. Πού και πόσες πιστώσεις έχουμε για τον τουρισμό, για επενδύσεις στον τουρισμό. Διότι είναι κρυμμένα σε διάφορα διευθυντικά ταμεία τα χρήματα και δεν είναι ορατά για χρηματοδότηση του τουρισμού. Αυτά δίδονται στα κράτη-μέλη που είναι υπεύθυνα για τη δαπάνηση και τη διοίκηση. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να δούμε πώς χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Επιπλέον, η πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις είναι πολύ πιο εύκολη για μεγάλες επιχειρήσεις παρά για μικρές. Αλλά το 90% των επιχειρήσεων του τουρισμού είναι μικρομεσαίες ε, και ιδιαίτερα μικρές επιχειρήσεις. Και αυτοί δημιουργούν, αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργούν και τις θέσεις εργασίας. Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα στις πιο διαφορετικές ευκαιρίες έχει ζητήσει μια ειδική γραμμή για τις δαπάνες για τον τουρισμό. Δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη γραμμή θα αυξήσει την ορατότητα. Από τη νέα χρηματοδοτική περίοδο υπάρχουν νέες διαδικασίες. Τα λεγόμενα λειτουργικά προγράμματα αποτελούν τη βάση για τη χρήση των πιστώσεων στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα για τις περιφέρειες. Και εδώ οπωσδήποτε θα προκύψουν θέματα και ελπίζω να δοθούν και σωστές απαντήσεις. Χαίρομαι λοιπόν για τη συζήτηση. Δυστυχώς ο αρμόδιος για την ειδική ομάδα τουρισμού, ο Ιστβαν Way, σήμερα δεν μπορεί να παρευρεθεί. Προβλέπουμε τρεις διαφορετικές συζητήσεις, κάθε ομιλητής μας έχει 5-6 λεπτά και σας παρακαλώ να τηρήσετε όλοι το χρόνο σας για να ολοκληρώσουμε ε, τη στιγμή που προβλέπετε. Πρώτος είναι ο κύριος Βούλφ από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Διαρθρωτικών Επενδύσεων. Κύριε Γούλφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Κυρίε ε, και κύριοι, να πω πως ε, βεβαίως ε, καλωσορίζουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα για τον τουρισμό να κάνω κάποιες ε, προκατακτικές παρατηρήσεις για τον τουρισμό και πώς τον βλέπουμε στην περιφερειακή πολιτική. Πρώτα απ' όλα η σημασία του τουρισμού ως ε, ένας σημαντικός οικονομικός κλάδος στις περιφέρειες και πρόκειται για μεγάλο κλάδο. Όπως ξέρετε είναι μεγαλύτερος από τον κλάδο των τροφίμων, ε, των αυτοκινήτων, των χημικών προϊόντων είναι γύρω στο 9 με 10% των εργαζομένων. Επιπλέον, έχει σημασία για να μπουν είναι η πρώτη φορά στην αγορά εργασίες και για τις επιχειρήσεις, όπως αναφέρατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά για τις μικρές επιχειρήσεις, νέους επιχειρηματίες ε, και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη και το πώς εργαζόμαστε εμείς στην προσέγγισή μας. Γιατί, γιατί δίνει ιδιαίτερη ε, βάση στην ε, ιστορία ενός τόπου τα πολιτιστικά του στοιχεία και την αηφορία βεβαίως για να διαφυλαχθούν όλα αυτά. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο νομίζω στην συζήτησή μας αφορά τον τουρισμό και τη συνεισφορά του στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή, πέρα από το ότι συνεισφέρει σε ανεπτυγμένες ε, περιοχές ε, και σε πρωτεύουσε, συχνά είναι οικονομικός παράγοντας σε λιγότερο ανεπτυγμένες και περιφερειακές ε, περιοχές, που ακριβώς εκεί πέρα ο καθοριστικός παράγον είναι η φύση. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, που συζητάτε σήμερα. Ο τουρισμός είναι κατά από άλλες ε, επικεφαλίδες ε, στην ε, περίοδο 2014-2017. Αν αναλύσουμε και ομαδοποιήσουμε τα ποσά, μιλάμε για 90 δισεκατομμύρια, 90 δισεκατομμύρια είναι διαθέσιμα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ως συγχρηματοδότηση για τις δημοσίες αρχές, αλλά Βεβαίως ε, και ως δάνεια και ως άλλοι τύποι επενδύσεων. Οπότε αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη μιλάμε για μεγαλύτερο ποσό. Αυτό αφορά τον τουρισμό αλλά υπάρχουν και επενδύσεις σε άλλους ε, τομείς. Προφανώς οι υποδομές των μεταφορών του περιβάλλοντος, οι ψηφιακές υποδομές που συνεισφέρουν στον τουρισμό και βεβαίως σε σχέση με τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οπότε το συνολικό ποσό είναι σαφώς μεγαλύτερο. από τα 9 αυτά δισεκατομμύρια. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και θέλουμε να φροντίσουμε ώστε να είναι διαθέσιμα αυτά τα κονδύλια μέσω των θεματικών στόχων που δεν αφορούν συγκεκριμένους κλάδους και να μπορούμε να διευκολύνουμε τον ε, τουρισμό όσον αφορά την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ή την ενίσχυση των μικρομισιών επιχειρήσεων ή την προστασία του περιβάλλοντος. Και σημασία έχει να γνωρίζουμε ότι το μισό περίπου ποσό αφορά την ενίσχυση και προστασία του περιβάλλοντος, ε, της πολιτικής κληρονομιάς και Κατόπιν έρχεται η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο στο πόσο ο τουρισμός μπορεί να ωφεληθεί από την εστίαση αυτής σε θεματικούς στόχους, αλλά και από την επιλογή των έργων, ε, έργα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να επεκτείνουν το τουριστικό προϊόν, να ενθαρρύνουν τον αηφόρο τουρισμό, θέλουμε κάποια καινοτόμο προσέγγιση, να επεκταθεί η βάση των πελατών, τα είδη του τουρισμού και θέλουμε να φροντίσουμε όλοι, όλα τα είδη του τουρισμού να συνεισφέρουν και θέλουμε επίσης ε, να ωφεληθεί ο τουρισμός από τις εξελίξεις ε, στον τομέα της ψηφιακής ατζέντα ε, του μάρκετινγκ, της προσβασιμότητας κτλ. Θα καταλήξω λέγοντας πως, ε, πως ξέρετε κάναμε μία αξιολόγηση εκ των υστέρων για την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης για τον πολιτισμό και τουρισμό και βγάλαμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρο και νομίζω πως το σημαντικότερο για τη σημερινή συζήτηση είναι πρώτον να ενσωματώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον πολιτισμό και τον τουρισμό στις ε, προοπτικές ε, και στην στρατηγική για την έξυπνη εξειδίκευση που δίνει βάρος στην ε, καινοτομία και στις επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες και στη διάσταση της αηφορίας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που προέκυψε από την αξιολόγηση είναι ότι πρέπει να περάσουμε από τις ε, επενδύσεις ε, σκληρές θα έλεγα υποδομές, δηλαδή ουσιαστικά από τα κτίρια στο να επενδύουμε στην ε, γνώση. Και βεβαίω να αναπτύξουμε περισσότερο τα επιχειρηματικά μοντέλα. Και βεβαίως αυτό το οποίο θεωρούμε ίσως ε, πρόκληση είναι το να ενημερώσουμε τις διαχειριστικές αρχές για το ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο ο τουρισμός και πώς μπορεί να υποστηριχθεί και να γίνει το ίδιο και για τους ε, εταίρους του τουρισμού. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ζιλ Τερτρέ από το γραφείο του Αντιπροέδρου της Κομισιόν του Γιουρκή Κατάινεν ο οποίος θα μας μιλήσει για τα μέσα της Ευρωπαϊκής, Κεντρικής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Σα ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μα δίνετε να βρισκόμαστε εδώ στην Επιτροπή σα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση γιατί πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τι ευκαιρίε που προκύπτουν από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, οι οποίε πρέπει να γίνουν απολύτω κατανοητέ. Προτού περάσω στις τη παρουσίασή μου, πρέπει καταρχά να πούμε ότι ε, οι ευκαιρίες του επενδυτικού αυτού σχεδίου δεν θα πρέπει να ειδωθούν ξεχωριστά από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Είναι απόλυτα συμβατές οι ευκαιρίες αυτές. Θέλουμε να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες και έχουμε και κάποια πρώτα παραδείγματα από έργα τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, αντίθετα με αυτό το οποίο πιστεύουν ορισμένοι, τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία δεν είναι μόνο μεγάλα έργα. Έχουμε καταρχάς τον τομέα που έχει να κάνει με την καινοτομία και τις υποδομές, έναν δεύτερο πυλώνα που έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους δύο αυτούς πυλώνες μπορούμε να κάνουμε χρηματοδοτήσεις προς τον τομέα του τουρισμού. Όσον αφορά τις υποδομές και την καινοτομία, αν δούμε το ΕΦΣΥ, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορούμε να συγκεράσουμε, να ομαδοποιήσουμε έργα, προκειμένου να έχουμε μία πλατφόρμα συνεπενδύσεων ουσιαστικά συνδυάζουμε δύο ή περισσότερα έργα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μπορεί να τα χρηματοδοτήσει πιο εύκολα. Θα έλεγα ότι είχαμε ασκήσει σημαντική πίεση σε χώρες όπως η Κύπρος ή η Ελλάδα, γιατί θεωρούμε ότι αυτού του είδους η χρηματοδοτική δομή, όπου θα μπορούσαμε δηλαδή να ομαδοποιήσουμε δυνάμει επενδυτές σε συγκεκριμένα έργα είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας και των υποδομών. Μπορούν να ομαδοποιηθούν κατά αυτόν τον τρόπο, να συνδυαστούν έργα και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για ορισμένα όργα, πιο συγκεκριμένα έργα στον τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε εδώ πέρα να έχουμε πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Το βασικό μήνυμα λοιπόν είναι ότι υπάρχουν οι ευκαιρίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με τα διαφορετικά ταμεία. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίσουμε τώρα προσπαθώντας να προωθήσουμε αυτές τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικής υποστήριξης. Χρειάζεται περαιτέρω τεχνική υποστήριξη προκειμένου να καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τα έργα αυτά και προκειμένου οι δικαιούχοι στον τουριστικό τομέα να καταλάβουν ότι υπάρχουν αυτές οι επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ακριβώς το λόγο με το επενδυτικό αυτό σχέδιο είπαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτός ο συμβουλευτικός κόμβος προκειμένου να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφές με τις δημόσιες αρχές, αλλά ακόμα και οι ιδιωτικοί φορείς, καταβάλλοντας ένα πολύ μικρό τέλος, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επενδυτικές συμβουλές μέσω του κόμβου αυτού. Την 1η Ιουνίου έχουμε και το τελευταίο εργαλείο για το επενδυτικό αυτό σχέδιο, η πύλη αυτή, ε, μια δημόσια ιστοσελίδα ουσιαστικά, όσον αφορά τις επενδύσεις που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΦΣΥ, όπου οποιοδήποτε φορέας έχει μια πολύ καλή ιδέα η οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΥ μπορεί να την υποβάλει σε αυτή την πύλη. Και δίνει τη δυνατότητα κατά αυτόν τον τρόπο ακόμα και στον τουριστικό κλάδο, ακόμα και σε φορείς από τον τουριστικό κλάδο να υποβάλουν τέτοιες επενδυτικές ιδέες μέσω της διαδικτυακής αυτής πύλης είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσελκύσουμε περισσότερε υποψηφιότητε από τον τουριστικό κλάδο, ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ορισμένε χώρε. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα τη οικονομία του. Αν λοιπόν γίνουν οι απαραίτητε επενδύσει στον κλάδο αυτό, θα καταφέρουν να έχουν και πολύ πιο θετικά αποτελέσματα για την οικονομία του. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ο κύριος Λουί Δεγκράντε Πασχουάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω πρώτος και ε, θέλω να σε ενημερώσω ότι η, Κλάιντ, η Κλάουδια Μοντέρο Δε Αγγιλάρ που πάντα ασχολείται με τα θέματα αυτά δυστυχώς ε, δεν μπορεί να είναι σήμερα παρούσα. Θα σας παρουσιάσω τις θέσεις της με τις οποίες συμφωνώ. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο, αλλά αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από αναδυόμενου προορισμού. Αν δεν ληφθούν μέτρα, θα μειωθεί το ποσοστό μας στην παγκόσμια αγορά. Το 2000 είχαμε το 51% του παγκόσμιου, της παγκόσμιας αγοράς. Τώρα είμαστε κάτω από 40. Και οι προβλέψεις είναι ότι θα υπάρξει περαιτέρω πτώση. Το 2030 προβλέπεται 31%. Άρα χρειαζόμαστε επενδύσεις για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Ο ευρωπαϊκός τομέας πρέπει να εφαρμόσει καινοτομίε, να προσαρμοστεί στις αλλαγές και τις τάσεις της αγοράς και να επενδύει συνέχεια στις υποδομές, την ε, συνδεσιμότητα, τη διαφήμιση, νέα προϊόντα, την ποιότητα των υπηρεσιών, νέες τεχνολογίες και βεβαίως την ψηφιοποίηση, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Βεβαίω είναι αρκετά σταθερή η τουριστική κίνηση κατά την κρίση, αλλά παρόλα αυτά διαπιστώνουμε ότι έχει μειωθεί οι, έχουν μειωθεί οι επενδύσεις κατά 15% γιατί έχουν μειωθεί οι δημόσιες επενδύσεις άρα δεν μπορούν να γίνουν οι βασικές επενδύσεις σε υποδομές ε, και την, την λειτουργία των μικρομεσαίων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τη μείωση των επενδύσεων και γι' αυτό έχουμε το σχέδιο επενδύσεων. Βεβαίως έχουμε το ΕΦΣΥ που θα κινητοποιήσει τουλάχιστον 315 δις. Αλλά με συνολικό προϋπολογισμό 450 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 14-20 τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν πολυετή προγράμματα. Ο τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για να υπάρξει ανάπτυξη και απασχόληση. Οπότε, ζωτικό είναι να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες ευκαιρίες και να, και, επαρκές, και να υπάρχει και ένα επαρκές ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτω ώστε να παραμείνουμε ο πρώτος τουριστικός προορισμός. Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Συγχαίρω την Κομισιόν για αυτή τη δυνατότητα επενδύσεων στον τουρισμό και για τις καλές πρακτικές εντός της Ένωσης. Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, τους οποίους ευχαριστώ στους ε, παρουσιαστές, τους οποίους ευχαριστώ. Πρώτη, ο προπολογισμό του κόσμου για το 2017 μειώθηκε κατά 50% και έχει πει ότι έχει αναλάβει δεσμεύσεις. Αλλά τι δεσμεύσεις όταν υπάρχουν τόσο δραστικές περικοπές, παρακαλώ, απαντήστε τι δυσχέρειες αντιμετωπίζετε για να μπορέσετε να χρηματοδοτηθείτε από το σχέδιο Juncker. Αναφερθήκατε ήδη σε αυτό, αλλά θα ήθελα να τους ζητήσω να μου απαντήσουν πιο συγκεκριμένα, για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα και συγκεκριμένα πώς τίθεται το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ. Jill Evans. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα σε αυτή την ειδική ομάδα. Αλλά επανερχόμεθα συνέχεια στα ίδια θέματα. Επενδύσεις. Σε πιο ήπιες υποδομές είπατε, στη γνώση και στον πολιτιστικό τουρισμό. Κάτι που με ανησυχεί στην έκθεση των υστέρων που είδα, ιδιαίτερα για την στήριξη από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, είδα ότι οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται στις αστικές περιοχές, όχι στην Ήπεθρο. Εγώ είμαι από την Ουαλία που είναι κυρίως ε, Ήπεθρος. Στην Ήπεθρο έχουμε λοιπόν λιγότερες επενδύσεις ε, σε υποδομές, ε, στις τηλεπικοινωνίες. Άρα ε, είναι σε μειονεκτική θέση η ύπεθρος. Θέτω λοιπόν το θέμα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και για τις μικρομεσαίες. Πώς μπορεί να τις βοηθήσει η Κομισιόν στις ε, συγχρηματοδοτήσεις τουριστικών προγραμμάτων. Αναφερθήκατε στο ΕΦΣΥ αλλά υπάρχουν ε, κάποιε αμοιβέ άμα θέλει κανεί να λάβει υπηρεσίε συμβούλων για να ζητήσει χρηματοδότηση. Υπάρχει κάποια στρατηγική να προσεγγίσουμε τι μικρομεσαίες, να του χορηγήσουμε αυτή τη στήριξη που χρειάζονται, την οικονομική βοήθεια, γιατί πολύ συχνά αγωνίζονται ούτω ή να τα βγάλουν πέρα ε, στη γενικότερη κατάσταση τη οικονομία. Υπάρχει τρόπο η Κομισιόν να κάνει πιο στοχευμένη βοήθεια προ τι μικρομεσαίες, να του βοηθήσουν να κάνουν αιτήσει είτε με μονομένε επιχειρήσει, είτε να συνεργαστούν κάποιε επιχειρήσει για να λάβουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Γένς, ο πρόεδρο, Γιάννη Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να τονώσουμε την ε, τουριστική δραστηριότητα, είναι να προωθήσουμε περαιτέρω την πολιτική συνοχής γιατί εκεί δαπανάται η μερίδα του λέοντος των ε, περιφερειακών ταμείων. Και το ελκυστικό στην πολιτική συνοχής είναι ότι εφαρμόζεται εκ των κάτω προς τα άνω. Αν μια περιφέρεια πει ότι στη δική μας αναπτυξιακή στρατηγική θέλουμε να συμπεριληφθεί ο τουρισμός, εδώ θέλουμε να στοχεύσουμε για να δημιουργήσουμε απασχόληση, ανάπτυξη, αυτή η στρατηγική θα είναι η βάση για τα προγράμματα του Περιφερειακού Ταμείου για αυτήν την περιφέρεια. Να αναφέρω ως παράδειγμα τη δική μου περιφέρεια, στη Σουηδία. Από τη δεκαετία του 90 έχουμε στοχεύσει περισσότερο στον τουρισμό για να έχουμε ανάπτυξη. Έχουμε χρησιμοποιήσει τα περιφερειακά ταμεία για να αναπτύξουμε προορισμούς, μέσω συνεργασίας επιχειρήσεων για να αναπτύξουν συγκεκριμένους προορισμούς, μέσω συγχρηματοδότησης από τις περιφέρειες και τους ΟΤΑ και το κοινωνικό ταμείο που είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Τέτοια προγράμματα είναι επίσης σημαντικά και βεβαίως οι μεταφορές για να μπορέσουν να μεταφερθούν οι πελάτες, αλλά πρέπει να υπάρχει πραγματική συμμετοχή των απλών ανθρώπων των εργαζομένων της περιοχής. Και αυτό μπορείς να το επιτύχεις μόνο αν τους κινητοποιείς από τη βάση. Και άκουσα εδώ στους διαδρόμους ότι θα πρέπει να καταργήσουμε την πολιτική συνοχή. Όχι, αντίστροφα. Αν θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε τον τουρισμό, πρέπει να βασιστούμε στην τοπική και περιφερειακή προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος. Τέιντρου Κλούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές. Νομίζω πως ε, είχαμε πολλές ε, συζητήσεις και συμφωνούμε ότι έχει μεγάλη σημασία για την απασχόληση ο τουρισμός, ειδικά στις περιφέρειες και για τους νέους. Ο κύριος Γουλφ ε, κοίταξε τα προηγούμενα επενδυτικά ταμεία και τα διδάγματα που αντλούμε για το επόμενο πρόγραμμα και υπάρχουν τρεις τομείς, ο πολιτιστικός τουρισμός, που είναι σημαντικός. Φαίνεται ότι δεν έχουμε τέτοια συνδυαστική σκέψη στην Ευρώπη. Κάθε περιφέρεια έχει την δικιά της κληρονομιά. Αλλά νομίζω από τη διαφημιστική σκοπιά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να προωθήσουμε την Ευρώπη ως ε, έναν χώρο πολιτιστικού τουρισμού. Γνωρίζω πως στην Ιρλανδία αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι κριτές για να διαλέξουν ποια θα είναι η πόλη, πολιτιστική πρωτεύουσα για το επόμενο έτος και θα είναι αυτό ένα τεράστιο πλέον έκτημα βεβαίως για την πόλη η οποία θα λάβει αυτό το βραβείο αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως μπορούμε να προωθήσουμε παραδείγματος χάρη τους δρόμους ε, του κρασιού, του φαγητού κτλ και βεβαίως ε, η έμφαση από τη σκληρή γνώση και τις σκληρές επενδύσεις τις πιο ήπιες ας πούμε γιατί οι υποδομές ε, χρειάζονται οπωσδήποτε στις ε, περιοχές της υπαίθρου και δεν πρέπει να ξεχνάμε τους δρόμους, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και αυτά θα είναι σημαντικά. Δεν θα υπάρχει τουρισμός διαφορετικά. για το θέμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τώρα. Το είχα κοιτάξει στην αρχή όταν ανέβηκε αρχές Ιουνίου, αλλά η ομαδοποίηση των έργων νομίζω μπορεί να βοηθήσει και πρέπει να το προωθήσουμε αυτό. Περιφερειές και χώρες δηλαδή να προωθήσουν διάφορα έργα. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε μετά αλλά το πώς θα μπορέσουν να υποφεληθούν οι επιχειρήσεις από την ομαδοποίηση αυτή, νομίζω θα είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ινές Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Δίνουμε βοήθειες σε διάφορους τομείς ε, και το αυτοκίνητο, για παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία, τους έχουμε δώσει πολύ περισσότερη βοήθεια. Ενώ για τον τουρισμό είμαστε αρκετά φιδωλοί. Θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις, να είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι. Βεβαίως καλό είναι, καλοδεχούμενη αυτή η χρηματοδότηση που δίνεται τώρα. Ξέρουμε ότι η Τράπεζα Επενδύσεων έχει δύο δυνατότητες, την φυσιολογική, ας πούμε, την παραδοσιακή και την άλλη που στα πλαίσια του σχεδίου Juncker ε, αναλαμβάνει περισσότερους κινδύνους στον τουρισμό. Όπως είπε και ο κύριος Χιλ Τέρτρε, έχουμε ξενοδοχεία, για παράδειγμα, που θα πρέπει να ανακαινήσουμε ή να δούμε πώς θα γίνουν ενεργειακά πιο αποδοτικά. ή πώς να βρούμε τρόπους στα πλαίσια μιας πιο φιλόδοξης προσέγγισης για τον τουρισμό, πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να πείσουμε την Τράπεζα Επενδύσεων να στοιχηματίσει περισσότερο σε σωστά προγράμματα, για παράδειγμα πολύ συγκεκριμένες σιδηροδρομικές γραμμές διαμεθοριακές που μπορούν να βοηθήσουν τον τουρισμό. Όπως για παράδειγμα ο διαπυρηναϊκός αυτός σιδηρόδρομος. Διότι το σχέδιο Juncker λέει ότι τα προγράμματα που θα επιδοτηθούν πρέπει να είναι επικερδή, αλλά πώς θα μετρήσουμε την κερδοφορία στην περίπτωση του τουρισμού. Σε άλλους τομείς, για παράδειγμα, είναι εύκολο να δεις ε, πότε είναι κερδοφόρα μία επένδυση. Αλλά εδώ πρέπει να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης. Πρέπει ας πούμε να δούμε τη δυνατότητα εξυγχρονισμού κάποιων ε, ε, υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και περιβαλλοντικά θέματα. Αυτή η δικτυακή πύλη τώρα, που προσπαθεί να φέρει σε, ιδέα, σε επαφή τις επιχειρήσεις με τους επενδυτές. Δηλαδή, πώς θα βοηθήσει για τον τουρισμό αυτή η δικτυακή πύλη να παρουσιάσουν, να διαφημίσουν τις ιδέες τους οι επιχειρηματίες και πώς όταν κάνουν κάτι τέτοιο προστατεύεται η ιδιοκτησία, προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των επιχειρήσεων αφού πρέπει να περιγράψουν τα προγράμματά τους θέλουμε να είναι ουσιώδη, καινούργια πρωτότυπα να προσφέρουν τη θέμα αξία. Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, γιατί πρέπει να τα κοινοποιήσουν όλα αυτά, να τα πούν στις τράπεζες κτλ. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε τα πνευματικά δικαιώματα. Έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα που να μα εξηγείτε πώ γίνονται αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα θα μιλήσω και εγώ έχω μια ερώτηση προς τον κύριο Γούλφ. Υπάρχει μια διαφορά με την χρηματοδοτική περίοδο μέχρι το 2014 και την επόμενη. Όταν μιλάμε για τα διαρθρωτικά ταμεία, της διαδικασίες και τις ε, προτεραιότητες, τι έχει αλλάξει και το θεωρείτε θετικό ή όχι. Και μετά μια άλλη ερώτηση για την συγχρηματοδότηση και την αποτελεσματικότητα ενός έργου. Στην ε, συζήτηση ακούσαμε ότι στο Γκέντιγκεν και το Ζόπελτ και το Ντάνσιχ εκεί στις τρεις αυτές πόλεις της ε, Πολωνίας θα χτιστεί ένα αεροδρόμιο 90 χιλιόμετρα από το παλιό αεροδρόμιο του Γκτάνσκ. Υποθέτω ότι είναι λόγω τουρισμού, αλλά ξέρουμε πως ένα περιφερειακό αεροδρόμιο δεν είναι ποτέ επικερδές μόνο με τον τουρισμό. Και πριν από μερικά χρόνια έκλεισε το αεροδρόμιο στο Ζαρμπρούκεν γιατί η Κομισιόν είπε ότι οι επιδοτήσεις για αυτό το αεροδρόμιο που απέχει 30 χιλιόμετρα από το Ζαρμπρούκεν και είναι και τα δύο λιματικά ε, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και χωρίς την επιδότηση έκλεισε. Πώς μπορείτε να κρίνετε και κρίνετε ε, όταν σας ζητάνε χρηματοδότηση για κάτι τέτοιο. Λέτε όχι, Κάτι άλλο, μεταξύ Βερολίνου και Ούζεντομ του νησιού υπάρχει μια πολύ καλή σύνδεση, αλλά βεβαίως η γέφυρα καταστράφηκε στον τελευταίο πόλεμο. Ξέρετε ότι είναι, πάνε πολλοί Βερολινέζοι για να κάνουν μπάνιο εκεί πέρα τα λοιπά και γενικώ έχει τουριστικό ενδιαφέρον. Αλλά αν δείτε το σιδηρόδρομο βλέπετε πως μόλις 4% των επιβατών πάνε με το τρένο. ή άλλοι πάνε με τα μάξι ή με άλλους τρόπους γιατί το τρένο κάνει τέσσερις ώρες ενώ εάν είχε γίνει η γέφυρα θα χρειαζόταν μόνο δύο ώρες. Με 100 εκατομμύρια για τη γέφυρα αυτή θα μπορούσαμε να συνδέσουμε πάρα πολύ καλά το Βερολίνο με το Ούζεντομ. Πώς το αξιολογείτε ή αν σας το ζήταγε ο σιδηρόδρομος θα δίνατε αυτά τα 100 εκατομμύρια από το Ταμείο Γιόνκερ για τη γέφυρα αυτή. Τι θα λέγατε ή τι θα με συμβουλεύατε εμένα για να πω στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Λοιπόν, κύριε Βούλφ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σχόλια. να πω το εξή. Κοιτάξτε, για τον αν είναι αποτελεσματικές οι επενδύσεις. Κανείς δεν θέλει να βρεθεί στην περίπτωση επενδύσεων που δεν είναι αποτελεσματικές ή υποκάθισαν κάτι άλλο. Και νομίζω το τονίσαμε όλοι. Σε σχέση με το αεροδρόμιο και την ερώτηση αυτή. Αυτό το οποίο θέλουμε γενικώ είναι να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια και επίσης να έχει μια στρατηγική περιφέρεια και να την έχει αναπτύξει σε συνεργασία με όλους τους υπόλοιπους ε, φορείς, ε, τις επιχειρήσεις ε, ιδιαίτερα και τους υπόλοιπους. Σε σχέση λοιπόν με οποιαδήποτε μεγάλη υποδομή θα κοιτάγαμε να είναι ενταγμένο σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο για την περιφέρεια και να έχει αξιολογηθεί σωστά ο οικονομικός αντίκτυπος. Και οπωσδήποτε δεν ε, θα θέλαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου θα επενδύαμε σε ένα δευτερεύον αεροδρόμιο χωρίς να έχει διασφαλιστεί το κύριο. Τώρα, για τις ε, επενδύσεις της ε, συνολικότερες ε, που νομίζω είναι αυτό το οποίο εννοείται με την γέφυρα και τα συνολικά ωφέλη. Κοιτάξτε, για την γέφυρα θα εξετάζαμε όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη κλαδικά αλλά συνολικά για να δούμε επίσης ε, τον συνολικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις και να τις συγκρίνουμε με έναν τρόπο ολοκληρωμένο. Δηλαδή θα κοιτούσαμε τα ωφέλη όχι μόνο όχι μεμονωμένα. Με ρωτήσετε ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της προηγούμενης και αυτής της ε, περίοδου. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι μόνο να υπάρχει μια αξιολόγηση των επενδύσεων όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, αλλά όπως είπαν και διάφοροι ομιλητές, θέλουμε να ενθαρρύνουμε την εμπλοκή των εταίρων στη λήψη των αποφάσεων. Αναφέρθηκε παραδείγματος χάρη η μαζική συμμετοχή και βεβαίως ε, και συμμετοχή των επιχειρήσεων. Έχουμε δηλαδή επενδύσεις ε, σε έργα τα οποία θα αναγνωρίζουν τις στρατηγικές ε, δυνάμεις και πλέον εκτήματα μιας περιφέρειας σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και βεβαίως να φροντίσουμε να υπάρχει ε, Ένα πολύ θετικός συνολικό αντίκτυπος. Κάποια πράγματα, κύριε Πρόεδρε, που θα ήθελα να αναφέρω. Με ενδιαφέρον άκουσα αυτό το ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις ε, περιοχές ε, της περιφέρειας ότι εξακολουθούν οι αστικέ περιοχέ να λαμβάνουν δυσανάλογο κομμάτι τη χρηματοδότηση. Δεν βλέπω κάποιο λόγο για να συμβαίνει αυτό, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να το δούμε με προσοχή, να δούμε γιατί οι περιοχές υπαίθρου δεν οργανώνονται έτσι ώστε να φροντίσουν οι επενδύσει να γίνονται εκεί. Και το άλλο βασικό θέμα που κοιτάμε είναι να φροντίσουμε να υπάρχει εμπλοκή των επιχειρήσεων και των άλλων φορέων. Ειδικά η φύση του τουρισμού που δίνει μεγάλη έμφαση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν ενδείκνεται οπωσδήποτε για εύκολη εμπλοκή των επιχειρήσεων. Και πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θα ακουστεί η φωνή των επιχειρήσεων να εμπλακούν στη διαδικασία και οι διαχειριστικές αρχές, οι υπεύθυνε να κάνουν μια σοβαρή συζήτηση. για το θέμα αυτό και την σχέση με τον τουρισμό. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίλ Τρέπε. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα μία ερώτηση σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για τη χρήση των ταμείων αυτών. Κοιτάξτε, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και μιλώντας με τους επιχειρηματίες, βλέπουμε το εξής. Πρώτον, υπάρχει ένα πρόβλημα γνώσης καταρχάς ότι φύστανται αυτά τα ταμεία. Να σας δώσω το παράδειγμα της, του κλάδου της έρευνας, όπου υποτίθεται ότι εκεί πέρα θα πρέπει να γνωρίσουν οι καλύτεροι ερευνητές ε, ποια είναι τα διαθέσιμα ταμεία παρόλα αυτά μιλώντα κανεί με καινοτόμε μικρομεσαίε επιχειρήσει, εντοπίζει ότι δεν γνωρίζουν καν ούτε και αυτές ποια είναι τα διαθέσιμα ταμεία για τη χρηματοδότηση τη έρευνα. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε και να προβάλλουμε περισσότερο τι ευκαιρίε που μπορούν να δώσουν τα ταμεία αυτά. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρόβλημα με την απλούστευση. Πρέπει να απλουστεύσουμε τι διαδικασίε, οι οποίε πολλέ φορέ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις κρατικές ενισχύσεις τα οποία πρέπει να επιληθούν. Όλα αυτά μας απασχολούν. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα της υπαίθρου. Πολύ θετική εντύπωση μας έκανε ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων υπάρχουν τελικά πολλά επενδυτικά έργα τα οποία προέρχονται από την Ήπεθρο. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στον αγροδιατροφικό τομέα. Εκεί έχουμε πολύ καλές επενδυτικές προτάσεις. και πολύ σημαντικά προϊόντα που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Ευρώπης και υπάρχει πραγματικά εκεί πέρα ένα πολύ σημαντικό δυναμικό. Να σας δώσω δύο παραδείγματα από το ΕΦΣΥ. Επενδύσαμε στην περιοχή της Νορμανδίας, στη Γαλλία, μια επιχείρηση που προθύνει μια καινοτόμα μέθοδο παραγωγής βουτύρου και μάλιστα η επιχείρηση αυτή έχει δημιουργήσει στην πόλη στην οποία βρίσκεται πολλές θέσεις απασχόλησης και κατάφερε κατά αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση να προχωρήσει σε πιο καινοτόμες μορφές παραγωγής. Ένα άλλο παράδειγμα, και μάλιστα αυτό είναι το πρώτο σχέδιο το οποίο κάναμε στην Ελλάδα που έχει να κάνει με το ελαιόλαδο, παραγωγή ελαιολάδου στην Κρήτη. Αν μπορούσαμε λοιπόν τέτοια θετικά παραδείγματα να τα προωθήσουμε περισσότερο, θα μπορούσαν να εμπλακούν και άλλε επιχειρήσει από άλλε περιοχέ. Νομίζω επίσης ότι πολύ σημαντικές ευκαιρίες μπορούν να προκύψουν από την ομαδοποίηση και το συνδυασμό διαφορετικών επενδυτικών έργων. Ξέρω ότι πολλές φορές παρουσιάζονται προβλήματα με ένα και μόνο επενδυτικό έργο. Πολλοί μπορεί να φοβούνται ότι ενδεχομένως να προκύψουν πολλά προβλήματα αν ομαδοποιήσουμε πολύ περισσότερα επενδυτικά έργα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το προσπαθήσουμε. λαμβάνοντα υπόψη επίσης και το περιορισμένο προσωπικό τη Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνουν οι άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε κάθε περιοχή ξεχωριστά. Ακριβώς επειδή όμως έχουμε αυτές τις επενδυτικές πλατφόρμες, μπορούμε ακριβώς να συγκεράσουμε πολλά διαφορετικά προγράμματα. Για παράδειγμα, στην περιοχή Ile France της Γαλλίας έχουμε τράπεζες, τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο το οποίο μπορεί στη συνέχεια να δοθεί με τη μορφή χρηματοδότησης στους ιδιοκτήτες ε, κατοικιών, σπιτιών και μάλιστα έχουν απευθυνθεί συνολικά σε 40.000 40.000 ε, ιδιοκτήτες ακριβώς για να γίνει μια ανακαίνιση των σπιτιών αυτών. Τώρα, δεν αποφασίσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα επενδυτικά σχέδια. Είναι ανεξάρτητη η ε, Επιτροπή η οποία αποφασίζει για τα ποια έργα θα πρέπει να επιλεγούν. Από τεχνική και οικονομική πλευρά πρέπει να είναι βιώσιμα. Αυτό είναι το κριτήριο. Δεν μπορώ να σα δώσω λοιπόν εγώ μία απάντηση για την επιλεξιμότητα των ε, έργων. Απλώ λέμε ότι οι επιχειρηματίε θα πρέπει να έρχονται όλο και περισσότερο σε επαφή με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών για να δουν τελικά αν μπορούν όντω να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά του έργα, να έχουν το σωστό προφίλ ή θα μπορούσαν να βρεθούν εναλλακτικέ μορφέ χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να κάνουμε τη δεύτερη συζήτηση για τη χρήση των ε, ενωσιακών ε, επενδύσεων από τα διεθνωτικά ταμεία. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Κοράτσα από τη Γενική Διεύθυνση GROW. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την πρόσκλησή σας. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα COSME βασίζεται όχι μόνο στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων, δηλαδή θέλει να προωθήσει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων, αλλά και τον τουρισμό. Για τη γενική μας διεύθυνση, ο τουρισμός έχει στρατηγική σημασία γιατί έχει πολλές επιπτώσεις και σε άλλους τομείς όπως οι κατασκευές, οι μεταφορές, η μόδα, τα προϊόντα πολυτελείας και ο αγροτροφημικός τομέας. Και υπάρχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης στον τομέα αυτό. Με βάση κάποιες προβλέψεις θεωρείται ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έως 500.000 νέες θέσεις εργασίας το χρόνο για την επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό θέλουμε να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Έχουμε ορισμένες προτεραιότητες. Πρέπει να στηρίξουμε τις προσπάθειες κατάρτισης, διότι οι ανάγκες του κλάδου δεν καλύπτονται. Τα προσόντα των εργαζομένων δεν είναι επαρκή του εργατικού δυναμικού. Επίσης για την ψηφιοποίηση, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες της ψηφιακή επανάστασης. Επίσης διεθνοποίηση, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών για περισσότερη ανάπτυξη και επίσης διαφήμιση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν πιο πολύ την ε, διαφήμιση των τουριστικών των προορισμών. Τα τελευταία χρόνια ο προπολισμός του κόσμου είναι 8 με 9 εκατομμύρια ευρώ, όχι πολύ μεγάλο ποσό, και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει περικοπές. Όμως ο προπολισμός του κόσμου μπορεί να παίξει ρόλο μόχλευσης για άλλους προπολογισμού, για την κατάρτιση για παράδειγμα. Το 2017 προβλέπουμε 800.000 ευρώ που θα προσθεθούν στα 4 εκατομμύρια του έρασμο ΣΥΝ. για να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου με τις διάφορες σχολές ε, και άλλους οργανισμούς κατάρτισης. Για να έχει το ειδικευμένο προσωπικό που θέλει ο κλάδος και για να μπορούν και οι νέοι να κάνουν ε, επισκέψεις ε, κατάρτιση σε άλλες χώρες και έτσι να αυξήσουμε τις δυνατότητες καταπολέμησης της πολύ ψηλή ενεργείας των νέων, ιδιαίτερα στον Νότο. Επίσης, ένα ταμείο για κοινή διαφήμιση, 3 εκατομμύρια του κόσμου, για να προσελκύσουμε και χρηματοδοτήσεις από άλλες γενικές διευθύνσεις και ιδίως των ε, περιφερειών και από τον κλάδο για να έχουμε πιο αποτελεσματική διαφήμιση στις τρίτες χώρες ο πρόεδρος Γιούνκερ ανέγγειλε ότι το 2018 θα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρονιά του τουρισμού σε συνδυασμό με την Κίνα. Άρα θα κάνουμε πολλές ε, δραστηριότητες ε, ευαισθητοποίησης στην Κίνα για να γνωρίσουν την Ευρώπη οι Κινέζοι. Τα επόμενα 15 χρόνια οι τουρίστες από την Ασία θα αυξηθούν κατά 500%. Έτσι λοιπόν θα επιχειρήσουμε με τους δικούς μας πόρους να συντονίσουμε τις προσπάθειες του κλάδου, τις άλλες προσπάθειες της Ένωσης και των κρατών μελών για να προσελκύσουμε περισσότερους Κινέζους τουρίστες. Να μόνο μερικά παραδείγματα για το πώς αξιοποιούμε τον προπλογισμό του κόσμου. Επίσης υπογραμμίζω ότι η Επίτροπος Μπινκόφσκα ανήγγειλε ενώπιόν σας ότι θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για να ε, προωθήσουμε τις ε, συνεργασίες μεταξύ του προϋπολογισμού μας και του κλάδου του πολιτιστικού και δημιουργικού τουρισμού μέσω πιλωτικών προγραμμάτων μαζί με τον ορίζοντα 2020 για την ψηφιοποίηση του μουσείου, ε, εικονική πραγματικότητα σε αριολικούς χώρους, άλλες δυνατότητες για να αξιοποιήσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και το 18, όπως ξέρετε, θα είναι και χρόνος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τέλος, στις 27 Σεπτεμβρίου, μαζί με την οργάνωση Next Tour έχουμε μία εκδήλωση με την επίτροπό μου, την ε, κυρία Μπενκόφσκα, για να συζητήσουμε με τις περιφέρειες και τους εκπροσώπους του κλάδου πώς θα εφαρμόσουμε το σχέδιο Juncker, πώς θα αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διαφροντικά ταμεία για να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα τουρισμού στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΦΙΟΥΣ ειδίκευσης και εξυγχρονισμού του κλάδου και στις 29 Νοεμβρίου θα έχουμε μια εκδήλωση για να παρουσιάσουμε τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης τουρισμός και ε, πολιτιστική και δημιουργική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Οικονόμου, από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που περιλάβατε και τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ μεταξύ των ομιλητών. Έχω έρθει να σας ενημερώσω για τις πρωτοβουλίες ε, και τις δράσεις που έχουμε αναλάβει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας και Θαλάσσης, το οποίο λεγόταν απλά Ταμείο Αλληλείας στο παρελθόν. Τώρα πλέον που λέγεται και Θαλάσσιο Ταμείο, έχουμε τις γενικότερες πτυχές της θαλάσσιας πολιτικής που απασχολούν τη γενική μας διεύθυνση πέραν από την Αλία. Και το κοιτάμε αυτό στο πλαίσιο της ε, γαλάζιας ανάπτυξης ε, και οικονομίας που περιλαμβάνει ε, ουσιαστικά και τον τουρισμό, τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό που είναι μία από τις μεγαλύτερες δραστηριότητες της λεγόμενης οικονομίας και εκπροσωπεί το 1 τρίτο, όπως είπαμε, της ε, θαλάσσιας οικονομίας. Ε, οι μεγαλύτερες προκλήσεις αναφέρθηκαν ήδη, η εποχικότητα, ανταγωνισμός από ανταγωνιστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως οι αλλαγές στα μοτίβο του τουρισμού, στις επενδύσεις, ε, το είπαν οι ομιλητές ειδικά με την κρίση, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Το 2014 λοιπόν υιοθετήσαμε μια στρατηγική για περισσότερη ανάπτυξη και δουλειέ ε, στον παράκτιο τουρισμό και έχουμε κάποιες δράσεις, οι οποίες παρακολουθούμε 13 στον αριθμό και οι Κομισιόν και οι τοπικές αρχές και τα κράτη-μέλη. Τι κάνουμε λοιπόν με τα λεφτά του ταμείου αυτού. Θα ξεκινήσω με τις πιο ήπιες δράσεις και μετά θα περάσω στις πιο ουσιαστικές ξεκινήσαμε με τον λεγόμενο πανευρωπαϊκό διάλογο για τον κλάδο της κρουαζιέρας, ένα πολύ δυναμικό κλάδο και όπως ξέρετε το Μάρτιο του 2015 συναντήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γύρω από τον κλάδο και μπορέσαμε έτσι να συζητήσουμε, να αναζητήσουμε κάποιες λύσεις και να προωθήσουμε νέες αγορές. Μετά ακολούθησε ο περιφερεια... ακολούθησαν οι περιφερειακοί η Μεσόγειος, η Βαλτική και θα συνεχίσουμε. Και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ε, της κάθε περιφέρειας. Και έρχομαι τώρα στις μελέτες. Έχουμε κινήσει διάφορες ε, μελέτες, ειδικά στον κλάδο του θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού και τις ε, καινοτόμες στρατηγικές για τις παράκτιες περιοχές Σημαντικά όλα αυτά για τους ενδιαφερόμενους γιατί μπορούν έτσι να ξεκινήσουν την στρατηγική τους να βρουν νέες αγορές και τρόπους προώθησης των προϊόντων τους. Και μετά, μιλώντας για προϊόντα, οι θεματικές και πολιτιστικές διαδρομές είναι πολύ της μόδας τώρα. Είναι μια νέα προοπτική που βλέπουμε στον τουρισμό και έχουμε απευθύνει μια πρόσκληση για να έρθουν διάφορες προτάσεις για πολιτιστικές διαδρομές στην Ευρώπη. Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον παρά τον μικρό προπολογισμό και αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τις προτάσεις που λάβαμε με την προκήρυξη αυτή. Και έχουμε προγραμματίσει επίσης φέτος με κάπως πιο ουσιαστικό προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο την δημιουργία διαδρομών στον ναυτικό τουρισμό. Και πάλι αναμένουμε ενδιαφέρον από τον κλάδο γιατί έτσι θα επιτραπεί η προώθηση του κομματιού αυτού του τουρισμού που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για πολλές περιφερειές στην Ευρώπη. Νομίζω επίσης πως οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ναυτική και πολιτιστική κληρονομιά που έχει τόσο μεγάλη σημασία στην Ευρώπη και υπάρχει και ευρωπαϊκό έτος που έρχεται για την πολιτιστική κληρονομιά το 2018 Οπότε αναπτύσσουμε διάφορες δράσεις. Βεβαίως, τώρα, περνώντας τα πιο σοβαρά που ξεκινήσαμε φέτος, είχαμε τις ε, προκηρύξεις ε, που αφορούν τις γαλάζιες λεγόμενες, που είναι τρεις τον αριθμό υπερκήρυξη για τις γαλάζιες ε, σταδιοδρομίες, για νέες προοπτικές για τους επιστήμονες εκείνους ε, που εμπλέκονται στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Μετά έχουμε τα γαλάζια εργαστήρια τα λεγόμενα, για τα καινοτόμα εργαστήρια και τους νέους επιστήμονες ε, που όπως πολλοί ανέφεραν πρέπει να προωθήσουμε για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω τη συγκεκριμένη πτυχή του ταμείου μας που συνδέει απευθείας την αλληλεία με τον τουρισμό, γιατί και στο παρελθόν, στον άξονα 4, είχαμε διάφορα έργα που προωθούσαν την ε, μετατροπή διαφόρων ελευτικών δραστηριοτήτων ε, και την επέκτασή του στον τουρισμό. Και στην περίοδο 2014-2020 προβλέπουμε γύρω στα 514 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις δραστηριότητες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη τοπικών δραστηριοτήτων όπως η προώθηση αλληλευτικών ταξιδιών, παρουσιάσεων σε σχολεία, το να πηγαίνει κόσμο σε αλληλευτικά σκάφη και έτσι θα υπάρχουν νέες προοπτικές για αυτές τις ε, κοινότητες. Ελπίζω λοιπόν να παρουσίασα τις διαφορετικές πτυχές ε, του πολιετούς ε, δημοσιονομικού πλαισίου και να σας έπεισα ότι κάνουμε αρκετά πράγματα για την προώθηση του παράκτηου και θαλάσσιου τουρισμού και να συνεισέφερα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και δεν έχουμε προσκαλέσει μόνο την Γενική Διεύθυνση ΜΑΡ, αλλά και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ο κύριος Καστελάνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια σύντομη παρουσίαση PowerPoint. Θα ήθελα να προβάλλω κάποιες διαφάνειες, αν είναι δυνατόν. Λειτουργεί πολύ ωραία λοιπόν. Καταρχάς σα. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλου. Θα ξεκινήσουμε με μια γενική παρουσίαση του όλου πλαισίου. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία θέλουμε να θίξουμε στα πλαίσια της πολιτικής μας. Ξέρετε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμα τον όρο τουρισμός στην Ήπεθρο, υπαίθριος τουρισμός, αλλά οτιδήποτε βλέπετε στη εφάνεια συνδέεται αυτή τη στιγμή με τουριστικές δραστηριότητες. Ο τουρισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και όλες αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στον τουριστικό κλάδο και υποστηρίζουν γενικότερα και τις παρεμφερείς δραστηριότητες. Ας μην ξεχνάμε για παράδειγμα πώς θα μπορούσε να προωθηθεί ο τουρισμός μέσω σημαντικών δραστηριοτήτων όπως είναι η γεωργία, η ε, ανακαίνιση γεωργικών μονάδων, η ανακαίνιση αναβάθμιση του ε, τοπίου της υπαίθρου κτλ. Αν δούμε την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και κάποια αριθμητικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από τον πίνακα που είχαμε παρακολούθηση για την προηγούμενη περίοδο, είχαμε δύο βασικά μέτρα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον γεωργικό τουρισμό, τον αγροτικό τουρισμό. Ο πρώτο είχε να κάνει με την ενθάρρυνση των τουριστικών δραστηριοτήτων, όπου χρηματοδοτήσαμε περίπου 20.000 έργα, που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη μικρών υποδομών, καθώς επίσης και υποδομών αναψυχής, είχαν να κάνουν ακόμα και με την ανάπτυξη εμπορική προώθηση τουριστικών υπηρεσιών στην Ήπεθρο. Επενδύσαμε πάνω από μισό δισεκατομμύριο ευρώ, όπου είχαμε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση στη συνέχεια και φτάσαμε περίπου τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε έπειτα και μία διαφοροποίηση εδώ πέρα σε σχέση με τις ε, καθαρά γεωργικές δραστηριότητες, όπως είπε και ο στάδελφος από την DG Mare, περίπου 0,20 δισεκατομμύρια δαπανίσαμε γι' αυτό και καταφέραμε να έχουμε περίπου 8.000 δικαιούχους, κυρίως ε, από τις αγροτικές περιοχές και αναφερόμαστε το κυρίως σε αγρότες. Επίσης, προωθήσαμε και συγκεκριμένες δραστηριότητες από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Ας δούμε τώρα πώς έχει ε, η κατάσταση για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Βλέπετε εδώ πέρα μια γραφική παράσταση όπου ουσιαστικά βλέπετε την κατανομή του συνολικού προπολογισμού. Συμπεριλαμβάνεται εδώ πέρα και η εθνική συγχρηματοδότηση βάσει συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Οι τουριστικές δραστηριότητες ανήκουν στην προτεραιότητα παριθμών 6, προώθηση δηλαδή κοινωνικής ενσωμάτωσης και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων πέρα από τη γεωργία και βλέπετε εδώ πέρα ότι προβλέπεται περίπου ένα 15% του συνολικού προπολογισμού για αυτές τις δραστηριότητες. Συμμετέχουν όμως και χρηματοδοτικά και υπόλοιπε προτεραιότητες ή μπορεί να έχουμε χρηματοδοτική υποστήριξη και από τις υπόλοιπε προτεραιότητες. Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσουν ε, τα προγράμματα αυτά και τα ταμεία οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα αυτά καθεαυτά. Βλέπετε εδώ πέρα πώς κατανέμεται ο προϋπολογισμός στα βασικά μέτρα που έχουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Πρωτικής Ανάπτυξης με γαλάζιο. Βλέπετε τους τομείς αυτούς που μπορούν να συνάδουν περισσότερα στον τομέα του τουρισμού, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων, η προώθηση μικρών επιχειρήσεων, νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, βασικές υπηρεσίες ανανέωση των υποδομών, ανανέωση και αναβάθμιση διαφόρων περιοχών της υπαίθρου ή χωριών. Βλέπετε στρατηγικής bottom-up από τη βάση προς τα πάνω όσον αφορά την τοπική ανάπτυξη και έχουμε ακόμα και την προσέγγιση αυτή που εμπλέκει περισσότερο τις τοπικές κοινότητες όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα περισσότερο και ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία. Μα δίνεται επίση η δυνατότητα μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτική Ανάπτυξη να προωθήσουμε κάποιου τοπικού φορεί τη υπαίθρου για να αναπτυχθούν περισσότερο στον τουριστικό τομέα και χρηματοδοτούμε επίση ακόμα και πιλωτικά προγράμματα ή προγράμματα που βρίσκονται σε φάση δοκιμή. Και προσπαθούμε επίση να χρηματοδοτήσουμε και διάφορα προγράμματα παροχής συμβουλών ή ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε όλοι να υποφεληθούμε από τη γνώση που έχουν συγκεκριμένοι φορείς. Τώρα, ποιες επιχειρήσεις, ποια προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα μέσα αυτά. Βλέπετε εδώ πέρα έναν κατάλογο των πιο βασικών προγραμμάτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν Αναφέρομαι σε αυτά γιατί αναφέρθηκαν σε αυτά και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Η δυνατότητα δηλαδή να στηρίξουμε χρηματοδοτικά επενδύσει σε ευρυζωνικά δίκτυα ή σε υπηρεσίε πληροφορική όσον αφορά πάντα την ύπεθρο. Μπορούμε να έχουμε ακόμα και κάποιες επιχειρήσεις start-up στον τομέα του τουρισμού, καλύτερη συνεργασία μεταξύ φορέων που ήδη αναπτύσσονται στον τομέα του τουρισμού και το καθεξής. Όλα αυτά τα ζητήματα τα κάλυψα στις προηγούμενε διαφάνειες. Προσπαθούμε εδώ πέρα, όπως βλέπετε, να υποστηρίξουμε κυρίως όχι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στη διαφάνεια αυτή βλέπετε κάτι το οποίο εμεί κρίνουμε ω αρκετά σημαντικό προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα στο τέλο τη ε, περίοδου προγραμματισμού. Ξεκινάμε πρώτα με μία ανάλυση των πραγματικών αναγκών. Λέμε στι ε, αρχέ διαχείριση ότι θα πρέπει καταρχά να μα πούνε τι θέλουν να πετύχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και προκειμένου να επιτευχθούν τα αποτελέσματα αυτά χρειαζόμαστε συγκεκριμένες στρατηγικές. Θέλουμε επίσης συνέργειες και συμπληρωματικότητα με άλλα ταμεία. Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη δεν λειτουργεί από μόνο του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αποτελεσματικό, αποτελεσματικά να διασυνδέεται με τα υπόλοιπα ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταβάλει πολύ σημαντικέ προσπάθειε στα πλαίσια τη νέα περίοδου προγραμματισμού για να αυξήσει την συμπληρωματικότητα. Θέλουμε επίσης να προσανατολίσουμε περισσότερο τη στρατηγική μας σε απτά αποτελέσματα, σε πραγματικές επιδόσεις και θέλουμε και έναν ενισχυμένο διάλογο, καθώς επίσης και την πρόθεση εταιρικών σχέσεων, προκειμένου να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε με έναν απτό διάλογο με, τους, με τις του επιχειρήσεις, τους φορείς σε επίπεδο υπαίθρου στις ε, αγροτικές περιοχές. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις και τώρα η Deirdre Λούμ. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε και νωρίτερα ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ε, γεωργικές περιοχές, με τις περιοχές της υπαίθρου. Γιατί όντως ε, έχουμε πολλά που μπορούμε να κάνουμε εδώ. και ιδιαίτερα αυτά που μας είπαν ε, οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης ΜΑΡΕ για τον τουρισμό στις παράκτης περιοχές είναι πολύ ενδιαφέροντα. Οι 14 ε, δράσεις που ανέφερε ο κύριος Οικονόμου μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς θα τις εφαρμόσετε γιατί υπάρχει τόση πληροφόρηση και υπάρχουν τόσες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης που είναι σημαντικό να έχουμε μια επισκόπηση για το πώς εφαρμόζονται οι δράσεις αυτές και πώς αξιολογούνται μετά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ο τουρισμός μπορεί να φέρει πολλή απασχόληση στην Ήπεθρο μέσω αεροδρομίων κτλ. Όλα αυτά για την γαλάζια ανάπτυξη και ο παράκτης τουρισμός, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό για πολλές περιοχές μας που περιέχουν παραλίες και ακτές. Κύριε, Digicrow, κύριε εκπρόσωπε της DigiGrow, κυρίως ε, που μιλήσατε για την κατάρτιση και την ψηφιοποίηση, είπατε ότι δεν υπάρχει ειδικευμένο προσωπικό γιατί η ψηφιοποίηση θα γίνει πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις που στο παρελθόν μπορεί να μην ε, ασχολιόντουσαν με τέτοιους τομείς. Δεν θεωρούν ότι χρειάζονται τεχνική γνώση, αλλά είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ανδεχόμενους ε, πελάτες τους. Σημαντικό λοιπόν η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. για να βοηθήσουμε συνολικά τον τουρισμό, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η προσπάθεια τονισμού αυτής της πλευράς και όλοι οι φορείς που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση το Σεπτέμβριο θα τα ξανασυζητήσουν όλα αυτά. Και ο εκπρόσωπος της ε, DG Agri, βέβαια, οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι παράγουν ε, τρόφιμα. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Έτσι διαπιστώσαμε τι ακριβώς γίνεται, πώς συνδέονται όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στην προσπάθεια όλοι αυτοί που θα μπορούσαν να λάβουν χρηματοδότηση να γνωρίζουν τις πηγές χρηματοδότησης. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Για τον τομέα της αλίας μπορείτε να μας αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα που επιτύχατε αυτήν την διαφοροποίηση για να επιτύχετε χρηματοδότηση. Τι συγκεκριμένα επιτύχατε, τι μπορείτε να κάνετε περαιτέρω. Δεύτερη ερώτηση. Τα προγράμματα αλληλείας είπατε ότι είναι και για τις ε, λίμνες, τις εσωτερικές λίμνες. Τι ποσοστό έχετε δαπανίσει για την αλληλεία στις λίμνες. Είπατε πως δεν είναι μόνο για τη θαλάσσια αλληλεία. Ε, Κάτι άλλο. Είναι γνωστό ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν και διάφορα μονοπάτια που περνάνε μέσα από χωράφια. Αλλά και δρόμοι. Και διαπίστωσα ότι αυτοί οι δρόμοι μέσα από, το, μέσα από τα χωράφια ορισμένε φορέ έχουν όριο ταχύτητα 70 χιλιόμετρα. Αυτά πια δεν είναι μονοπάτια, μονοπάτια είναι κανονική δρόμη και έφυγα από εκεί. Αυτό ο συνδυασμό με ενδιαφέρει δηλαδή πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτούς τους δρόμους αν θέλουμε ε, αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές να περνάνε από πόλεις μου υπόθηκε ότι ε, εάν θέλουμε να το κάνουμε έτσι για να χρηματοδοτήσουμε και ε, λωρίδες για ποδηλάτες δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί ο πολιτιστικός τουρισμός δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ε, λωρίδες για ε, ποδηλάτες. Πώς μπορούμε όμως να χρηματοδοτήσουμε και αυτές τις λωρίδες. Παρακαλώ. Κύριε Κοράτσα, θέλετε να ξεκινήσετε. Σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τις πολιτιστικές αυτές διαδρομές, ναι, μας ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα αυτό και γι' αυτό συνεργαζόμαστε με την DG Mare, την DG Agri, την DG Regio. Και ξέρετε ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει ένα Ινστιτούτο όσον αφορά τις πολιτιστικές αυτές διαδρομές και ασχολείται επίσης και η ίδια η UNESCO. Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι έχουμε κάποια τουριστικά προϊόντα τα οποία είναι διεθνικά. και είναι σημαντικό να αντιλαμβάνεται ο κόσμο τα προϊόντα αυτά, όχι αναγκαστικά ως περιφερειακά εθνικά προϊόντα, αλλά ως ευρωπαϊκά πολιτιστικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεργαστούμε για το ζήτημα αυτό, για τη διαχείριση του προπολογισμού κόσμε, αλλά και τη διαχείριση των υπόλοιπων ταμείων, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να προωθήσουμε όλες αυτές τις πολιτιστικές διαδρομές χρησιμοποιώντας το δίκτυο της UNESCO και συνειδητοποιώντας παράλληλα ποιες είναι οι θετικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο για τοπική οικονομία. Ένα ακόμα παράδειγμα το οποίο σας έδωσα ήταν να χρησιμοποιήσουμε κάποιες διαδικτυακές πύλες όπως αυτή της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης προκειμένου οι νέοι να μπορούν να κάνουν άσκηση κατάρτιση σε ξενοδοχεία για παράδειγμα. Ένας νέος, για παράδειγμα, ο οποίος έχει παρακολουθεί ένα περίοδο κατάρτισης στην Αυστρία το χειμώνα, θα μπορούσε να συνεχίσει την κατάρτισή του αυτή, την περίοδο άσκησης, σε μια άλλη περιοχή της Νότιας Ευρώπης, για παράδειγμα στην Ισπανία ή στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά να δώσω και το λόγο στους συναδέλφους που έχουν σίγουρα πολλά πράγματα να πούνε και αυτοί. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα το θέμα που αφορά τις ε, δράσεις ε, σε σχέση με την ανακοίνωση. Πράγματι αναφέρθηκα σε 14 τέτοιες. μπορώ να σας πω πως στις περισσότερες από αυτές έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Τα παραδείγματα που έδωσα ήταν ε, μεταξύ αυτών των δράσεων που περιέχονται στην ανακοίνωση. Παραδείγματο χάρη είναι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε τώρα για τον ε, ναυτικό τουρισμό, ο διάλογος για την κρουαζιέρα επίσης. Υπήρχε μια δράση για να κλείσουμε το κενό για τα οικονομικά δεδομένα του τουρισμού που είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορούν να προγραμματίσουν τις μελλοντικέ τους δραστηριότητες. Ε, μπορούμε λοιπόν με τη Eurostat να αναπτύξουμε μια καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων και προσπαθούμε να δούμε πώς θα έχουμε καλύτερα δεδομένα. Επίσης, οι μελέτες που ανέφερα. Επίσης, ε, περιγράφονται στην ανακοίνωση, παραδείγματος χάρη, η συνδεσιμότητα των νησιών. Επίσης ε, είχαμε προβλέψει έναν οδηγό χρηματοδότησης για τον παράκτιο και ναυτικό τουρισμό και θαλάσσιο τουρισμό, μέρος του γενικότερου οδηγού των συναδέλφων στην DG Είχαμε ένα παράρτημα που δίναμε συγκεκριμένα παραδείγματα για παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό. Και με περηφάνεια να πω πως ε, έχουμε προβλέψει και άλλες δράσεις ε, στην ανακοίνωση αυτή ειδικά καθώς έχουμε και αυτό το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς που ανέφερα. Τώρα, προβλέπουμε το 2018 να επανέλθουμε με τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης, οπότε η απάντησή μου στο ερώτημα πότε θα αξιολογήσουμε και τι αναφορά θα δώσουμε για τα αποτελέσματα. Σκοπεύουμε να κάνουμε μια εκδήλωση υψηλού επίπεδου και να σας αναφέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Μετά, να έρθω στο δικό σας το ερώτημα για την αλληλεία και συγκεκριμένα έργα. Να σας πω πως στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, 2007-2014, είχαμε χρηματοδοτήσει γύρω στα 409 εκατομμύρια ευρώ σε 12.000 τοπικά έργα για αυτή την μετατροπή και μετάβαση από την αλληλεία στον τουρισμό σε 21 κρατη Ένα καλό παράδειγμα θετικό παράδειγμα, γιατί εγώ δεν ήμουν καν σε αυτή τη γενική διεύθυνση τότε, αλλά ε, διαβάζω τι εκθέσεις των συναδέλφων, είναι στην Ελλάδα, όπου είχαν αναπτύξει τέτοιες δραστηριότητες, ε, μετέτρεψαν ε, σκάφη σε μουσεία, προωθούσαν αλιευτικές εκδρομές και ταξίδια και προωθούσαν και την πολιτιστική κληρονομιά της αλληλείας ως κομμάτι της τοπικής ε, παράδοσης. Εκεί έχουμε λοιπόν καλά παραδείγματα, αλλά υπάρχουν και πολλά, αλλά όπως είπα σε 21 κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω πως ήταν μια πρωτοβουλία που είχε θερμή υποδοχή και νομίζω ξοδέψαμε σωστά τα λεφτά. Σας ευχαριστώ. Γι' αυτό θα μιλήσετε τώρα ή μετά. Αλλιώς θα ακούσουμε τον κύριο Καστελάνο. Λοιπόν, ο κύριος Καστελάνο. Um, it's, it's on. Λειτουργεί. Με ακούτε. Πολύ ωραία. Ακούσαμε μία ερώτηση για την εμπλοκή των δυνάμει δικαιούχων στις πληροφορίες που δίνονται από το Ταμείο για τη Χρηματοδότηση. Ναι, μα ακριβώς για αυτό το λόγο είπαμε ότι πρέπει να έχουμε εταιρικέ σχέσεις και την εμπλοκή των ενδιαφερομένων σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού, του κύκλου προγραμματισμού, από, την, από το σχεδιασμό των προγραμμάτων μέχρι την ε, φάση της ε, υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Αυτό γίνεται μέσω της Επιτροπής ε, Παρακολούθησης και Εποπτείας στις διάφορες περιφέρειες των κρατών μελών, όπου προσπαθούμε να εμπλέξουμε τους δυνάμει δικαιούχους στην όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να ενημερώνονται περισσότερο και αυτοί για τη δυνατότητα χρηματοδότησης. Ο συνδυασμός τώρα διαφορετικών επενδυτικών έργων Ξέρετε ότι Αναφερόμαστε εδώ πέρα σε κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει πολύ συχνά και στο παρελθόν. Πού σταματάει το αστικό, πού ξεκινούν δραστηριότητε υπαίθρου. Έγινε μία απόπειρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν και έχουμε θετικά αποτελέσματα προωθώντα διάφορε μορφέ συμπληρωματικότητα στη χρήση των ταμείων αυτών. Το είπαν και οι συνάδελφοι αυτό. Να σε κάθε περιφέρεια τελικά να αποφασίσει με τρόπο διορατικό και συνεκτικό ποια είναι η καλύτερη για αυτήν λύση και αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τελικά το ένα ή το άλλο ταμείο. Αλλά πέρα από την χωριστή αυτή επιλογή δίνεται πλέον και δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών ταμείων, συνδυασμού διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων για ένα επενδυτικό έργο. Το κάναμε αυτό και στα πλαίσια των συμφωνιών εταιρική σχέση, προσπαθήσαμε να μαδοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα ταμεία για να προωθήσουμε κάθε δυνατότητα συμπληρωματικότητα. Και στι διαφάνειέ μου αναφέρθηκα ακριβώ στο ζήτημα αυτό. Διάλογο και συντονισμό. Ο διάλογο και ο συντονισμό θα πρέπει να γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Και θα πρέπει να εμπλέκεται βέβαια και η δημόσια διοίκηση προκειμένου να ενημερώνονται όλοι για τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αν όμως οι άνθρωποι δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, αν δεν υπάρχει ένας πιο διάλογος μεταξύ των φορέων χρηματοδότησης και των δικαιούχων, δεν πρόκειται να καταφέρουμε να προωθήσουμε αυτή τη μέθοδο χρηματοδότησης. Ευχαριστώ και περνάμε στον τελευταίο γύρο. Θα ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Νούνιες από το Next Tour και τον κύριο Μπόντορ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, με ακούτε. Ωραία. Η κυρία Νούνιες. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, κυρίε και κύριοι, με μεγάλη χαρά εκπροσωπώ την Next Tour για να σας αναφέρω ποιες είναι οι ποια είναι η οπτική γωνιά των περιφερειών. Εμείς εκπροσωπούμε 31 αρχές που ασχολούνται με τον τουρισμό, τον αηφόρο τουρισμό στις περιφέρειες, οπότε είμαστε ειδικοί στην χωροταξία, ανάπτυξη προϊόντων και στην προώθηση και εμπλεκόμαστε στην διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις επενδύσεις στις περιφέρειες. Οπότε αυτό εξηγεί ότι τώρα μία από τις τέσσερις ε, δραστηριότητε μας είναι η έξυπνη χρησιμοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον τουρισμό. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πρακτικά μπορούμε να διακρίνουμε τον ρόλο των περιφερειών ε, ανάλογα με το αν ε, είναι δικαιούχοι ή δωρητές και βεβαίως μετά ανταγωνίζονται με τους ε, άλλους ε, ενδιαφερόμενους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάποιους από τους στόχους ε, και τα προγράμματα είναι συμβατά. Π.χ. το ΕΤΠΑ και ορίζοντας 2020. Σύμφωνα με τα εργαλεία αναζήτησης, 49 περιφέρειες έχουν περιλάβει τον τουρισμό αμέσως ή εμέσως στην στρατηγική τους και βεβαίως γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα σήμανσης, καθώς ο οριζόντιος αυτός κλάδος συνδέεται και έχει πολύ πιο ε, σοβαρό αντίκτυπο σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρισμό και την αναψυχή όπως θα προσπαθήσω να σας δείξω. ο τουρισμός είναι βασικός κλάδος της ε, οικονομίας ε, και γράφεται στα περιφερειακά αυτά προγράμματα, τότε συγκεκριμένα μέτρα, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προβλέπεται. Και είναι σημαντικό βεβαίως για όλα αυτά να περιλάβουν την λέξη τουρισμό στα επιχειρησιακά προγράμματα. Οπότε πώς γίνεται αυτό. Ας δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη Σκωτία ο τουρισμός ε, ανήκει στο χαρτοφυλάκιο τουρισμού, πολιτισμού και εξωτερικών υποθέσεων ε, που περιλαμβάνει και έναν ε, Υπουργό εξωτερικών και ευρωπαϊκών υποθέσεων. Έχουμε λοιπόν τον οργανισμό, το Visit Scotland. Με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, μιλάτε λίγο γρήγορα. Ο οργανισμός, ο Visit Scotland, είναι αρμόδιος με την προώθηση της ε, Σκοτίας ε, και είχε συντάξει το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι διαχειριστής ενός προγράμματος ε, του ΕΤΠΑ η πρωτοβουλία αυτή λοιπόν στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ολόκληρη την Σκοτία για να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες από το εξωτερικό μέσω ενός ε, συνδυασμού ψηφιακών διάβλων, στήριξης ε, του κλάδου και διεθνών εκδηλώσεων. Τώρα, η αλληλεπίδραση με τον τουρισμό φαίνεται γενικά στην Σκοτία, στους κλάδους, ε, τον, ε, στον δημιουργικό κλάδο, τον κλάδο της εστίασης, ε, την ναυτιλία και τον τουρισμό. Τώρα βλέπουμε το παράδειγμα της Ανδαλουσίας. Παραδοσιακός προορισμός της Νότιας Ευρώπης που τώρα ανασχεδιάζει την στρατηγική της και περνάει σε μια πιο καινοτόμο προσέγγιση και πάει σε μια έξυπνη εξειδικευσή. Μάλιστα. Το ΕΣΥΦ και ειδικότερα το ΕΤΠΑ και RDF ε, προχωρούν στην στρατηγική από τώρα μέχρι το 2020, δηλαδή να υπάρξει αηφορία και ανταγωνιστικότητα του τουρισμού στην Ανταλουσία ως ένα στρατηγικό τομέα για την περιφερειακή οικονομία, δημιουργία θέσεων εργασία και την οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω στήριξη των επιχειρήσεων, ανακαίνιση και αναζωογόνηση του κλάδου, με την πρόθεση της Ανταλουσίας ως ενός προορισμού αριστείας και πρόθεση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Τα αποτελέσματα λοιπόν που αναμένουν είναι να έχουν ανταγωνιστικό τουριστικό κλάδο και να καταπολεμήσουν την εποχικότητα. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχει μια στρατηγική έξυπνη εξειδίκευση με τον τουρισμό, γιατί όπω λένε χρειάζεται έρευνα και ανάπτυξη και καινοτομία για να προσαρμοστεί στις αλλαγές της αγοράς που είναι βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου. Και κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι στην Ανταλουσία έχουν την δική τους προτεραιότητα για τον τουρισμό που λέγεται «Ενίσχυση της ε, Ανδαλουσίας ε, ως κέντρο αναψυχής ε, και πολιτισμού» και έτσι συνδέεται με καινοτόμα προϊόντα, προσβασιμότητα, πολιτισμό και βεβαίως συνέργεια με τις άλλες προτεραιότητες στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Λίγα λόγια τώρα για τις διασυνδέσεις τουρισμού με τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα. Στην Βαλένθια συνδυάζουν το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ για να στηρίξουν το Ινστιτούτο για τις τεχνολογίες του τουρισμού, προβλέπουν προγράμματα διαβίου κατάρτισης και καταπολέμησης ανεργίας των νέων. Στην Τοσκάνη το ΕΤΠΑ προσφέρει κάποια κουπόνια για την ε, καινοτομία στις επιχειρήσεις αρκεί να υπάρχει κάποια καινοτομία στους προορισμούς και αυτό γίνεται με το να γίνει ρητή αναφορά στην Ευρωπαϊκή ε, Ανακοίνωση της Κομισιόν 2010. Στη γερμανόφωνη κοινότητα του Βελγίου έχουμε το ΕΤΠΑ και το EARDF για να προσελκύσουν νέες ε, επενδύσεις και στην Κορνουάλη συνδυάζουν τρία ταμεία και το Ταμείο της Αλληλείας που αναφέρθηκε πριν μεταξύ αυτών και συνδέουν και τον τουρισμό. Καταλήγοντας λοιπόν, δεδομένης τη μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και στο μέτρο του δυνατού, ε, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη πρόσβασιμότητα και ορατότητα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αντιληφθούν καλύτερα τον ρόλο τους και τις ευκαιρίες που έχουν με τους στόχους του προγράμματος και τους στόχους που πρέπει να επιτύχουν. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, ειδικά όσον αφορά την προσαρμογή στις δραστηριότητες του τουρισμού. Θεωρούν πως ο τουρισμός ε, ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα της αγοράς σε αντίθεση με τον προσανατολισμό στην αναψυχή που υπήρχε παλαιότερα. Πρέπει να μην υπάρχει μεγάλη περιπλοκότητα, αναφέρθηκε αυτό, για να υπάρχει και ευελιξία. Θεωρούμε πως ε, η μεγαλύτερη ευελιξία θα αντιμετωπίσει καλύτερα την φύση του τουρισμού, καθώς πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις, ε, εποχιακές ε, και υπάρχει και ψηφιοποίηση πλέον και αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή όπως ήδη είπαν οι Γενικές Διευθύνσεις Ρέγγιο και Γκρο. Επίσης με περισσότερη λογοδοσία. Θεωρούμε πως πρέπει να έχουμε σωστά στοιχεία για τον αντίκτυπο άμεσο και έμεσο του τουρισμού. Συγκεκριμένες πρακτικές πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα μεταξύ του Στρατηγικού Ταμείου Επενδύσεων και των λοιπόν προγραμμάτων. με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για να στηριχθούν περισσότερο οι ανάγκε τη αγορά. και εδώ πέρα πιστεύουμε πώ η δημιουργία διεθνού τουριστικού προϊόντος απαιτεί ακριβώς την συνέχεια αυτών των επενδύσεων. Οπότε όλες οι φάσεις ανάπτυξης του προϊόντος θα πρέπει να έχουν ένα μακροπρόθεσμο όραμα και τέλος αναφέρθηκε ήδη περισσότερη επικοινωνία, περισσότερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Να πω πως η Nextour είναι μέλος του Μανιφέστου για τον τουρισμό, την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας και θεωρούν πως είναι μια πλατφόρμα για να φέρουμε καλύτερα τα μέσα αυτά πιο κοντά στον χρηματοοικονομικό κλάδο και βεβαίως σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Γι' αυτό ακριβώς χαιρόμαστε που συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση που ανέφερε η κυρία Κοράτσα τον Σεπτέμβριο με την Επιτροπή των Περιφερειών και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Είστε όλοι προσκεκλημένοι για να συζητήσουμε πώς θα ενθαρρύνουμε περαιτέρω τις έξυπνες επενδύσεις στον τουρισμό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much also for... Ευχαριστώ πολύ και για το ότι προσαρμόσατε την ταχύτητα της ομιλίας σας. Και τώρα ο Άνταμ Μπόντορ από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατών. Ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω ως αντιπρόεδρος της ομάδας για το Μανιφέστο για τον τουρισμό που κατήρτισε ένα θαυμάσιο κείμενο με πολλές προτάσεις για τον τουρισμό. Εκπροσωπώ την Ομοσπονδία Ποδηλατών που περιέχει είναι ο οργανισμός ο ευρύτερος που εκπροσωπεί ενώσεις όπου συμμετέχουν 500.000 ε, πολίτες. Έχω επίσης εργαστεί το παρθόν και σε, για μια αρχή διαχειριστική και γι' αυτό επιτρέψτε μου να είμαι λίγο πιο επικριτικός για τη χρήση των ε, ενωσιακών πόρων. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ε, για τα ποσά που έχουμε στη διάθεσή μας και κατά πόσο είναι προσιλωμένη η χρήση τους. Ε, ποιες είναι οι διαστάσεις των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται και πόσο βιώσιμα είναι αυτά τα προγράμματα, τα συγχρηματοδοτούμενα. Πρώτα απ' όλα, η χρηματοδότηση, το ύψος. Ε, βέβαια, καλά, ποτέ δεν είναι επαρκή τα ποσά. Όλοι οι κλάδοι θέλουν περισσότερα αλλά ειλικρινά. Ο τουρισμός ε, παρέχει το 9,7 του ΑΕΠ της Ένωσης. Και ο κύριος Χόφερ είπε ότι υπάρχουν περίπου 9 δις για τον τουρισμό από τα διαθροτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής. 9 δις. Δεν είναι απόλυτα σαφές. Μέσω ποιων προγραμμάτων θα λάβουμε αυτές τις χρηματοδοτήσεις αν είμαι ένας ξενοδόχος ας πούμε, αν έχω μια μικρή επιχείρηση στην Ήπεθρο, πού θα τα βρω αυτά τα εννιά δις, πού είναι διαθέσιμα για να αναπτύξω την μικρομεσαία μου επιχείρηση. Αν είμαι υπεύθυνο για ένα ιστότοπο για τον τουρισμό, πού θα πάρω χρηματοδότηση, μέσω της περιφέρειάς μου, πού ακριβώς είναι. Και αν θέλεις να κάνεις κάτι περισσότερο διεθνικό, μέσω του Interreg για παράδειγμα, δεν υπάρχουν πόροι. Ζητήσαμε για πόρους από το Interreg για την Κεντρική Ευρώπη και τη Βορειοδυτική. Είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την προσέγγιση που δεν είναι κλαδική. Και μου απάντησαν όχι άλλα τουριστικά προγράμματα. Σαφώς. Θέλουν να έχουν γενικότερα προγράμματα για την ε, βοήθεια προς μικρομεσαίες, αλλά όχι ειδικά τουριστικά. Τι πάει να πει όχι συγκεκριμένους κλάδους. Άρα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή ένα συγκεκριμένο κλάδο όπως ο τουρισμός δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριε Κοράτσα είπατε ότι έχετε 8-9 εκατομμύρια στο κόσμο. Ξέρω ότι κάνετε ό,τι μπορείτε για να δαπανίσετε με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα χρήματα για τον τουρισμό. Κοιτάξτε ένας κλάδος που είναι 9,7 του ΑΕΠ, του ενωσιακού ΑΕΠ. Και τι τους δίνουμε? 8-9 εκατομμύρια το χρόνο. Και περικόπτονται. Ξέρω ότι οι ευρωβουλευτές θέλουν να υπάρξει ειδική γραμμή για να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Αλλά είναι απόλυτα ανεπαρκές απόλυτα ανεπαρκές. Κάνουν ό,τι μπορούν. Αλλά τι να κάνουν, θαύματα με 9 εκατομμύρια. Πρέπει να αλλάξουν αυτά τα πράγματα, να είμαι σαφής. Και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο πρέπει να είναι πιο εμφανές πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί κανείς από αυτά τα 8-9, αλλά πρέπει να αυξηθούν κιόλα. Τώρα για την ποδηλασία δημιουργήσαμε ένα παρατηρητήριο. Ελέγξαμε όλα τα λειτουργικά προγράμματα. Είναι κάποιες εκατοντάδε, πολλή δουλειά, για να δούμε τι περιέχουν για την ποδηλασία. Αυτό πρέπει να γίνει και για τον τουριστικό κλάδο. Ποια λειτουργικά προγράμματα αναφέρονται εκπεφρασμένα στην ποδηλασία. Για την περίοδο 7-13 μόνο αν υπήρχε σαφής αναφορά στην ποδηλασία οι περιφέρειες επένδυσαν για αυτά, για κάποιες λωρίδες ή με άλλο τρόπο. Αν δεν υπήρχαν αναφορές δεν γινόταν. Κάναμε μια καμπάνια και μέσω των μελών μας. 1,6% των πόρων ε, των μεταφορών πάνε για την ποδηλασία, ενώ είναι 7,5% τα ταξίδια με ποδήλατο αλλά πρέπει να γίνει κάτι παρόμοιο για τον τουρισμό γενικότερα. Να κάνει μια καμπάνια για να καταστεί σαφές πού είναι οι πόροι για τον τουρισμό. Πώς αξιοποιούνται τώρα οι πόροι. Γιατί δεν αρκεί να υπάρχουν πόροι, πρέπει και να αξιοποιούνται σωστά. Όταν ήμουν σε μια διαχειριστική αρχή, εξεπλάγιν, από το ότι τα πριν που παίρναμε στο τέλος του χρόνου εξαρτώνται από το πόσα δαπανούσαμε. Αν ήσουν στο ιδιωτικό τομέα, δεν, παίρνατε, δεν παίρνεις στον ιδιωτικό τομέα μπόνους αν έχεις ξοδέψει περισσότερα από τους πόρους επιχείρησης. Άλλα κριτήρια θα μπορούσαν να ήταν, για παράδειγμα, πόσες περισσότερες διανεκτηρεύσεις υπήρξαν, πόση περισσότερη ανάπτυξη υπήρξε μέσω των τουριστικών προγραμμάτων. Αυτές είναι οι σωστές παράμετροι. Το ύψος των επιδοτήσεων πρέπει να συνδέεται με το αποτέλεσμα, όχι απλώς με το ποσό που δαπανάτε. Ξέρω ότι το ελεκτικό συνέδριο λέει ότι το κόστος δεν είναι το κύριο. Βλέπετε εδώ μια φωτογραφία ενός συναδέλφου που διαχειριζόταν ένα ε, μικρών διαστάσεων πρόγραμμα 400.000 ευρώ και βλέπετε πόσο γραφειοκρατία. Νομίζω ότι οι μικρομεσαίες, εάν έχουν μια καλή ιδέα, δεν πρόκειται να ζητήσουν επιδότηση γιατί είναι τόσο κοπιαστικό, έχει τόση γραφειοκρατία. Μήπως θα μπορούσαν να υπάρχουν για παράδειγμα κατά αποκοπήν πληρωμές με βάση την αρχή ε, ε, σωστή αξιοποίηση των πόρων. Τώρα διαστάσεις. Με εξέπληξε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι για τη στήριξη μικρομεσαίων από τις Βρυξέλλες. Για παράδειγμα μέσω των, ε, του ΕΦΣΙ και από το Κόσμε. Δεν ξέρω μήπως έχω λάθος ε, αντίληψη, έχω μιλήσει στις λάθος μικρομεσαίες. Αλλά όπως τα βλέπω εγώ, είναι σχεδόν αδύνατο να έρθουν στις Βρυξέλλες, να δουν πώς λειτουργεί το σύστημα και να λάβουν χρηματοδότηση. Νομίζω ότι η προσέγγιση του προγράμματος LEADER, όπου η διαχειριστική αρχή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο χορηγεί την πληροφόρηση να μάθει ένας ξενοδόχος τώρα πώς να ζητήσει χρηματοδότηση από τα διαφθορτικά και επενδυτικά ταμεία ή ένα site πώς να εφαρμόσει τέτοια προγράμματα είναι πολύ δύσκολο. Θα σας έλεγα οι πόροι αυτοί να αξιοποιούνται για ευρωπαϊκών διαστάσεων προγράμματα, δημιουργώντας δέσμες προγραμμάτων, συνδέοντας προγράμματα, συνδυάζοντας σε τοπικό επίπεδο πρέπει να στηριχθούν από τους πόρους που χορηγούνται ακριβώς σε τοπικούς φορείς προς διαχείριση και βιωσιμότητα. Είμαστε οργανώσεις ε, ποδηλατών, άρα μας ενδιαφέρει βιωσιμότητα. Ποτέ δεν είδα να είναι κριτήριο επιλογής αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σημαντικό για ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει τώρα περισσότερο είναι η οικονομική βιωσιμότητα. Ορισμένα νοσιακά προγράμματα θέλουν εντελώ καινούριε και πρωτότυπε ιδέε ιδιαίτερα τα διαμεθοριακά προγράμματα. Δεν μα ενδιαφέρει τι θα γίνει άμα λήξει το πρόγραμμα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Αν δείτε πώς λειτουργούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και πώς επιτυγχάνουν και πώς διατηρούν τη θέση τους στις αγορές, αυτό πρέπει να μας δείξει πώς να λειτουργούμε. Δεν μπορούμε κάθε δύο-τρία χρόνια να δημιουργούμε νέες μάρκες. Είναι πολύ επικίνδυνο. Θα ήθελα να επιδιώξουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις με στρατηγικούς εταίρους, με στρατηγικά προγράμματα. Αντί κάθε λίγο να ξεκινάμε με νέες ιδέες, νέες επιχειρήσεις, νέες μάρκες. Αυτό θα ήταν πιο βιώσιμο και θα παίζαν πολύ περισσότερο οι επενδύσεις μας. Συγγνώμη αν ήμουν λιγάκι γκρινιάρης. Ελπίζω να ε, σας έδωσα τροφή για συζήτηση και είμαι στη διάθεσή σας για όλα αυτά τα θέματα να σας πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε. Σας έχουμε καλέσει εδώ πέρα, όχι μόνο για να μας πείτε τι καλά είναι τα ευρωπαϊκά έργα, αλλά να μας πείτε και τις αρνητικές ε, πτυχές. Και πράγματι έτσι έγινε και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα ίσως ακούσουμε και άλλες αρνητικές εμπειρίες, αλλά πρώτα απ' όλα ακούσουμε την Ιζαμπέλα Ντεμόντε. Ευχαριστώ. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά τις ομιλίες αυτές που ακούσαμε και να αφαιρθώ σε μια γενικότερη ιδέα στην αρχή. Αν δούμε λίγο τη στρατηγική που ακολουθείτε, νομίζω ότι τα κονδύλια αυτά, τα ταμεία αυτά, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε άμεση χρηματοδότηση γιατί οι πολιτικές μας πολύ συχνά είναι περιφερειακές πολιτικές. Αν θέλουμε όμως πραγματικά να παραμείνουμε ο πρώτος προορισμός από τουριστικής πλευράς, ε, τότε θα πρέπει να υπάρχει και ένα συντονισμός, έτσι δεν είναι, και να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο με μία φωνή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία άκουσα από τον κύριο Κοράτσα όσον αφορά το πρόγραμμα COSME, ότι προσπαθεί να καταβάλει τόσο σημαντικές προσπάθειες χρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κονδύλια COSME είναι πολύ σημαντικά και βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν απτά αποτελέσματα και ήδη αυξάνεται αυτή τη στιγμή η γνώση και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένας οδηγός για τη χρησιμοποίηση των ταμείων αυτών. Γιατί ξέρετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απευθυνόμαστε κυρίως, απαρτίζονται βασικά από επαγγελματίες οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς λειτουργούν αυτά τα ταμεία. Αν λοιπόν έχουμε ήδη κάποια πρώτα απτά αποτελέσματα από τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων επενδύσεων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για την προσέγγιση bottom-up, από τη βάση προς τα πάνω. Νομίζω επίση ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεκτική τοποθέτηση για κάποια ζητήματα. Αναφερθήκατε στην Κίνα και είπατε ότι θέλετε να προσελκύσουμε περισσότερους Κινέζους τουρίστες. Ε, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όχι μόνο τα αγγλικά, αλλά ενδεχομένω και την κινέζικη γλώσσα και να έχουμε μια πιο άμεση προσφορά, αν θέλετε, του τουριστικού προϊόντος και να μην απευθυνόμαστε μόνο σε μεγάλα γκρουπ Κινέζων που έρχονται, αλλά και σε μονομένους επισκέπτες. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να προωθήσουμε περισσότερο ακόμα και τις άμεσες πτήσεις από την Κίνα, γιατί μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε τελικά να αυξήσουμε την έλευση Κινέζων τουριστών από την Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δημιουργήσουμε επίσης περισσότερες ε, ευκαιρίες σε εθνικό επίπεδο. Και θα πρέπει βέβαια τα προϊόντα τα οποία προτείνουμε στον τουριστικό τομέα να ανταποκρίνονται περισσότερο στη ζήτηση. Και κάτι άλλο. Το ζήτημα της ε, προσβασιμότητας μεγαλύτερη προσβασιμότητα αλλά και ορατότητα και προβολή όσον αφορά τα επενδυτικά ταμεία και στα πλαίσια κάποιου ιστότοπου, κάποιας ιστοσελίδας, να μπορούμε δηλαδή να έχουμε άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Εγώ ίδια προσπάθησα να το κάνω αυτό και δεν ήταν πολύ εύκολο να καταφέρω να δω τη σελίδα αυτή στην οποία αναφερθήκατε. Νομίζω λοιπόν ότι για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αποθεληθούν από τα ταμεία αυτά, θα πρέπει ενδεχομένω να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα, ένα ιστότοπο, ο οποίος θα είναι πιο προσβάσιμος, προκειμένου να υπάρχει άμεση προσφορά πληροφοριών στον ενδιαφερόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές. Νομίζω συνοψίσατε αυτό το οποίο είπαμε, ότι δηλαδή υπάρχει κόσμος που μπορεί να ωφεληθεί από αυτή τη χρηματοδότηση και απορούν, ε, δεν ξέρουν πώς θα λάβουν τις πληροφορίες. Νομίζω είπατε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για το ότι δεν πρέπει να αλλάζουν τα προγράμματα τόσο συχνά για να μπορούν να μαθαίνουν τις πληροφορίες οι άνθρωποι και να μην εμφανίζεται κάθε τρεις και λίγο ένα νέο πρόγραμμα που ανακαλύπτει ξανά τον τροχό. Είπατε λοιπόν κάποια σημαντικά πράγματα. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Νούνιας. Ήταν πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπατε. Θα ήθελα να μάθω πόσες περιφέρειες εκπροσωπείτε. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν πορές πληροφορίες για το πώς μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ τους οι περιφέρειες ε, και είμαι σίγουρη πως ε, ε, αυτό ευνοεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην κάθε περιφέρεια. Αναφέρατε διάφορες περιφέρειες και το πώς χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το κόσμο για να τα χρησιμοποιήσουν. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν πόσες περιφέρειες εκπροσωπείτε και τι κάνουν όσον αφορά τον ε, διαμοιρασμό οι πληροφορίες. Λοιπόν, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες οι εμπειρίες σας και διευκρινίζουν ακριβώς ε, τα προβλήματα που και εμείς αντιμετωπίζουμε ε, εδώ και πολλά χρόνια. Από τότε που είμαστε 28 με όλες τις περιφέρειες, με την διαφορετικότητα και τον μεγάλο πλούτο. Πάντα θεωρούσαμε ότι ο τουρισμός ήταν ένας τομέας που υπέφερε από την επιτυχία του, διότι λειτουργούσε από μόνος του ως θαύμα. Δεν υπήρχε λόγος ε, δημοσίων επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όλοι θεωρούσαμε ότι έχει μια γενική δυναμική, δεν χρειάζεται ενίσχυση όπως άλλοι τομείς. Δεν χρειαζόταν ούτε καν να επενδύσουμε. Δεν θα πω περισσότερα για τις διαφορές ε, βορρά-νότου Ανατολής Δύσης, γιατί κουράζομαι να λέω τα ίδια. Γιατί ορισμένοι λένε ότι χρειάζονται επενδύσει, δεν λένε ότι όλα γίνονται από μόνα του. Να δούμε ποια είναι η δομή του τραπεζικού κλάδου. Μετά την ε, οικονομική κρίση, σε ορισμένα κράτη-μέλη, οι περιφερειακέ τράπεζε, τα ταμιευτήρια που είχαν υποχρέωση να έχουν και μια κοινωνική πολιτική, να βοηθούν τι ε, περιφέρειές τους, Εξαφανίστηκαν όλες αυτές τις τράπεζες γιατί έγιναν πολλές ε, συγχωνεύσεις τραπεζών. Τώρα δεν θα την περιγράψω γιατί αρρωσταίνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι μικρομεσαίες, επειδή ούτως ή άλλως ξέρετε ότι οι μισοί εργαζόμενοι που είναι άνεργοι χρειάστηκε να γίνουν ε, υποθετικά αυτοαπασχολούμενοι, καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί δεν μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο επίπεδό τους, στο οικονομικό τους επίπεδο. Μια μικρομεσαία βέβαια δεν αντιμετωπίζεται σωστά από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτές οι μεγάλες τράπεζες του ζητάει να συνενωθούν για να έχουν πολύ μεγαλύτερη διάσταση για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Αλλά αυτές οι μικρομεσαίες είναι ένα σημαντικό τμήμα του τουρισμού. Υπάρχουν ε, μεγάλα ξενοδοχεία, εντάξει, ε, έχουν αυτά τις αναγκαίες ε, διαστάσεις, αλλά οι μικρομεσαίες που όμως είναι υπεύθυνε για την οικονομική και κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Ίσως πρέπει να κάνουμε κάποια έκκληση με βάση αυτά που μας είπαν η κυρία Νούνιεθ και ο κύριος Μποντόρα ακριβώς για την εξέβρεση λύσεων, τρόπων για να αποκτήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με συγκεκριμένες αρχές, με συγκεκριμένες αξίες ευρωπαϊκές. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν δυνατότητες που χρησιμοποιούνται σε άλλα πλαίσια. Στον ορίζοντα 2020 οι επιχειρήσεις ε, έχουν 25% των αμέσων ε, εξόδων τους, των αμέσων δαπανών των, ε, να χρωματοδοτείτε χωρίς να τους ζητάνε τίποτα. Όπως είπε και ο αρμόδιος ε, των ποδηλατών, πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες που διατηρούν τους ευαίσθητους κοινωνικούς ιστούς σε περιοχές που υπάρχουν πολλά προβλήματα. Να βοηθήσουμε πως βοηθούμε τις start-up. Βοηθάμε τις πιο σύγχρονες, τις πιο δημιουργικές. Εδώ λέμε ναι, να αναλάβουμε κινδύνους, να χάσουμε και λεφτά. Αλλά στον κλάδο του τουρισμού όλα πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται. Ναι. Παρθενογένεση. Άρα ως πορίσματα αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας συζήτησης θα μπορούσαμε να πούμε σαφώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει τρόπους ούτω ώστε ένα τομέα που δημιουργεί τόσε θέσει απασχόληση, που δημιουργεί συνοχή, που δημιουργεί την ε, αντίληψη για το τι είναι Ευρώπη, τη μάρκα Ευρώπη, ένα τέτοιο τομέα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει βοήθεια, χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρξει ακριβώ χρηματοοικονομική δημιουργικότητα για να βοηθήσουμε όσο γίνεται τον κλάδο αυτό είναι από τους τομείς που με κάθε άποψη μπορεί να θεωρηθεί δημιουργικός και βοηθάει στη διατήρηση της πολυμορφίας, της διαφορετικότητας της ένωσής μας. Θα ζητούσα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια προσπάθεια για να αντιμετωπίσει με μια γενναιόδωρο τρόπο και με πιο δημιουργικό τρόπο ε, τον κλάδο αυτό, γιατί αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι λυπηρά. Ευχαριστώ και Ζήνε Ευχαριστώ, ευχαριστώ και για την παρουσίαση όσοι άκουσα βεβαίως, αλλά για τον τελευταίο μιλτή να ρωτήσω συγκεκριμένα. Είπατε πως θα πρέπει να μετρήσουμε με βάση την επιτυχία τη χρηματοδότησή μας. Να κάνω λοιπόν μία ερώτηση. Μα αν κάτι είναι επιτυχές, χρειάζεται οικονομική στήριξη, μήπως να πούμε ότι λειτουργεί από μόνο του. Δεν είναι ανάγκη να χρηματοδοτούμε και να επιδοτούμε μονίμως τα πάντα, ε, ειδικά αν είναι επιτυχημένα. Δεύτερον, είπατε πως υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία και τα ακούμε συνεχώς. Δεν τον θέμε ε, κάτι τέτοιο επί της αρχής να υπάρχει δηλαδή υπερβολική γραφειοκρατία που θα πρέπει να ξεπεράσει κάποιος για να λάβει τις επιδοτήσεις και τις αναγκαίες επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως ε, θέλουμε πάντα να αποφεύγουμε την κατάχρηση, να υπάρχουν αποδείξεις για τα πάντα. Δεν είναι απλό λοιπόν, το γνωρίζω. Συγκεκριμένα λοιπόν, τι σας ενοχλεί, ποιες συγκεκριμένες προτάσεις έχετε για την απλοποίηση. Συγκεκριμένα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Γιάννη Νίλσον. Ε, ευχαριστώ. Ο τελευταίο ομιλητής επιβεβαίωσε αυτό το οποίο είχα πει, πω. η ανάπτυξη του τουρισμού πρέπει να έχει μια εστίαση τοπική και περιφερειακή. Γι' αυτό ανέλαβα την πρωτοβουλία να ζητήσω μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όπου θα μιλάμε για τη σημασία του τουρισμού, για την περιφερειακή ανάπτυξη μαζί με την αρμόδια επιτροπή, την Ρέτζη και μας το λένε αυτό οι περιφέρειες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Γιατί εάν μια περιφέρεια κρίνει ότι είναι στρατηγικό ζήτημα πρέπει τότε να δημιουργήσουν τη γνώση, την εμπειρογνωμοσύνη, ένα σχέδιο για το πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός στην περιφερειά του. Αν μελετήσουμε τις 50 καλύτερες περιφέρειες στην Ευρώπη που εστιάζουν στον τουρισμό, μπορούμε να δούμε το τι έκαναν και επέτυχαν. Νομίζω πως μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα έτσι. Θα ήταν ε, πολύτιμο λοιπόν να δώσουμε λεφτά για αυτή την ε, εμπειρογνωμοσύνη. Μετά, για τη γραφειοκρατία στα ευρωπαϊκά έργα. Η εμπειρία μου είναι ότι ο κόσμος λέει ότι είναι πολύ γραφειοκρατικά, αλλά η διαφορά με τις μικρές επιχειρήσεις είναι ότι συνασπίζονται για να κάνουν ένα μεγαλύτερο έργο, πιθανώς σε συνεργασία με την περιφέρεια ή τον Δήμο και έτσι μειώνεται η γραφειοκρατία με το να συνασπίζονται όπως σας είπα και να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η περισσότερη γραφειοκρατία δεν δημιουργήθηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά από τα κράτη-μέλη. Οπότε στα κράτη-μέλη πρέπει να απευθυνθείτε και να τους πείτε να μειώσουν την ε, γραφειοκρατία. Γιατί εκεί χρειάζεται η απλοποίηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω κάτι και μπορείτε να απαντήσετε μετά κυρία Κοράτσα. Η κυρία Μπόντο είπε πως ε, ο τουρισμός ε, πλέον ε, δεν πρέπει να επιδοτείται και μετά μας είπε και η κυρία Μάισνερ μας είπε το ίδιο. Κοιτάξτε, υπάρχει ο ευρωπαϊκός αυτός δρόμος, ο 6 και ο 13 που πάει στον Δούναβη, στη Σερβία κτλ. Και είπε τώρα, για ποδηλατόδρομο μιλάμε, και είπε θα βάλουμε απλά κάτι νέες πινακίδες και θα έχουν και κάποια ρητά. κάτι πινακίδες που γράφανε πέρα από διάφορα ρητά, είχε και κάτι άλλες που λέγανε Nice You Bed Service. Ε, πρόκειται λοιπόν για πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί βεβαίω ξέρετε ότι ξοδεύουν πολύ περισσότερα λεφτά οι ποδηλάτες από έναν τουρίστα που έρχεται με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, Αν έρθουν π.χ. οι Πολωνοί και πούν ότι έχουμε 400 χιλιόμετρα δύο ποδηλατόδρομους, αλλά 10 χιλιόμετρα από αυτά ε, είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση που χρειάστηκα 3 ώρες για τρία χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν ανάγκη να λέμε ότι ο ποδηλατικός τουρισμός είναι επιτυχημένος, δεν χρειάζεται λεφτά. Μπορούμε στοχευμένα να ξοδεύουμε. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν, ε, γιατί είπατε τέρμα τώρα ο τουρισμός και δεν θα το χρηματοδοτούμε άλλο. Και τώρα τέλος για την ε, γραφειοκρατία. Στην Άιζενστατ που είχα πάει μου είπαν πως ο Δήμος ότι μπορούμε να ζητήσουμε, τους είπα μπορείτε να ζητήσετε ευρωπαϊκά κονδύλια. Και μου είπαν όχι είναι τόσο σπολικό πως δεν έχουμε τόσα λεφτά, προτιμούμε να το πληρώσουμε μόνοι μας. Δηλαδή, αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πάνε τα ευρωπαϊκά κονδύλια μόνο σε μεγάλες επιχειρήσεις. Ε, είναι άδικο αυτό και αντικοινωνικό. Και εδώ πέρα πρέπει να το σκεφτεί και η Κομισιόν αυτό. Τι θα κάνει. Δεν είναι δυνατόν οι μικροί δήμοι που χρειάζονται ακριβώς αυτή τα λεφτά να λένε δεν θα ασχοληθώ γιατί κοστίζει πάρα πολύ και οι μεγάλες επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόβλημα να υπομισθούν το κόστος να λαμβάνουν την επιδότηση και να έχουν ε, βγει και να έχουν κερδίσει πριν ξεκινήσουν καν. Αυτά θα ήθελα να μου απαντήσετε. Λοιπόν, η κυρία Νούνιες. Yes, thank you Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που ακούσαμε. 31 περιφέρειες εκπροσωπεί το δικό μου το δίκτυο και αυτό συνδέεται με 33 επίσης πανεπιστήμια καθώς επίσης και άλλα δίκτυα βιώσιμης, βιώσιμου τουρισμού. Ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές για το πώς επωφελείται ο τουρισμός από τα κοινοτικά κονδύλια. Το 2013 έγινε αυτό γιατί τότε έγινε και η διαπραγμάτευση του πρώτου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου και τότε είχαμε και τι συγκεκριμένε προτάσει όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ήταν δύσκολα τα πράγματα στην αρχή για τα μέλη μα, γιατί έπρεπε ουσιαστικά σε περιφερειακό επίπεδο οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να καταλάβουν πώς γίνεται η μετάβαση από το προηγούμενο MFF στο υφιστάμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και έπρεπε επίσης να δούνε πώς θα καταφέρουν να εντάξουν περισσότερο τουριστικές επενδύσεις. Και πολλές φορές μεταξύ των περιφερειών έπρεπε να ασκηθεί περισσότερη πίεση προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να εμπλέξουμε όλα τα μέλη μας στη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Εν μέρη τουλάχιστον κατάφεραν να καταλάβουν καλύτερα πώς λειτουργούν οι τεχνικές ιδιαιτερότητες χρηματοδότησης για το τουριστικό τομέα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε τώρα την εφαρμογή της χρηματοδότησης και γι' αυτό έχουμε εκδηλώσεις για την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών όπως το Σεπτέμβριο. Τον Ιανουάριο είχαμε μια στρογγυλή τράπεζα για ένα από τα θέματα αυτά. Ο κύριος Γουόλφ ήρθε και μας είπε τότε για το πόσες περιφέρειες συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά χρηματοδότησης και όταν απεύθυνα, με συγχωρείτε, το ζήτημα αυτό προς τους συμμετέχοντες, υπήρχαν ε, μόνο τα μέλη του δικού μου δικτύου τελικά που σήκωσαν το χέρι για να συμμετέχουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς απαραίτητες γνώσεις ακόμα. Πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλουν οι περιφέρειες για να μεγιστοποιήσουν τις επενδύσεις στον τουρισμό, χρειαζόμαστε πιο άμεση υποστήριξη και από τις Βρυξέλλες. Όχι επειδή ανθίσταται αυτή τη στιγμή ο τουρισμός ε, στην οικονομική κρίση. Δεν είναι ότι επειδή αντέχουμε σαν κλάδο στην οικονομική κρίση ότι δεν χρειαζόμαστε δηλαδή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όντως έχουμε καταφέρει να δώσουμε συγκεκριμένε πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα παραδείγματα από τις περιφέρειες και νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητούμε περισσότερο τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν μεγιστοποιήσει περισσότερο τις ευφυείς αυτές ευκαιρίες για την πρόθεση περισσότερο του τουρισμού, τουρισμού στα πλαίσια των περιφερειακών στρατηγικών. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε επίσης και ποιες είναι οι δαφικές επιπτώσεις από την πρόθεση του τουριστικού κλάδου. Ο κύριος Μποντόρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε δύο ερωτήματα. Πρώτον, για ποιο λόγο επενδύουμε δημόσια κονδύλια και για ποιο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η κυρία Μάισνερ και ένας ακόμα ευρωβουλευτής έθεσαν το ζήτημα αυτό. Πρώτον, γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός στην παγκόσμια αγορά τουριστικών υπηρεσιών. Η Ευρώπη βρισκόταν στην πρώτη θέση σε όλες τις πτυχές του τουρισμού. Τα πράγματα όμως τώρα αλλάζουν και ο ποδηλατικός τουρισμός δεν είναι πλέον μόνο ευρωπαϊκός, υπάρχουν και άλλες χώρες, άλλες περιοχές του κόσμου που επενδύουν στον κλάδο αυτό. Υπάρχουν και άλλες ήπειροι εκτός Ευρώπης που κάνουν επενδύσεις σε αυτόν τον ποδηλατικό τουρισμό. Πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική. Στα πλαίσια πάντως του τουρισμού υπάρχει μία ιδιαιτερότητα, ένα ζήτημα το οποίο δεν ομοιάζει με τα χαρακτηριστικά άλλων κλάδων. Στον τουρισμό οι επενδύσεις και οι δαπάνες γίνονται πολύ συχνά από διαφορετικούς φορείς σε σχέση με το κέρδος και τα πραγματικά ωφέλη. Για παράδειγμα, ο Μίχαελ Κράμερ αναφέρθηκε στους ποδηλατοδρόμους. Μία τοπική κυβέρνηση ας πούμε ότι χρηματοδοτεί ένα ποδηλατόδρομο. Και ενδεχομένως βέβαια οι όσοι χρησιμοποιούν το δρόμο αυτό να μην μείνουν καν στα ξενοδοχεία που βρίσκονται πάνω στο δρόμο αυτό σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα επωφεληθούν ενδεχομένως κάποιοι άλλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσοι βρίσκονται πάνω στον ποδηλατόδρομο αυτό, οι ίδιοι οι κατασκευές του ποδηλατόδρομου δεν καταφέρουν τελικά να αποφεληθούν. Έχουν κάνει τις δαπάνες για την επένδυση, άλλοι καρπώνονται τα κέρδη από την επένδυση αυτή. Αυτό γίνεται πολύ συχνά με τις δημόσιες επενδύσεις και τις επιτυχίες. Τώρα, πώς μπορεί να μειωθεί η γραφειοκρατία, ένα άλλο ζήτημα το οποίο τέθη. Δεν θα ήθελα να περάσω πολλές λεπτομέρειες τώρα. Αναφέρθηκα σε κάποιες ταξιδιωτικές δαπάνες. Αν για παράδειγμα κλείσω το εισιτήριο του αεροπλάνου του τρένου αρκετά νωρί, τότε πετυχαίνω και καλύτερη τιμή. Αν το κάνω τελευταία στιγμή, τότε πληρώνω τεράστια τιμή. Και τα δύο όμως είναι αποδεκτά και για τις διαχειριστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρκεί να έχω το εισιτήριο στο χέρι μου. Για ποιο λόγο να μην υπάρχει ένα καταποκοπήν ποσό. Για ποιο λόγο να μην γνωρίζουμε καλύτερα κάποιες ε, τυποποιημένες τιμές όσον αφορά ή πολλές φορές όσον αφορά και το ίδιο το προσωπικό. Σε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούμε πάρα πολλούς εργαζομένους μας οι οποίοι πρέπει να συμπληρώνουν όλες αυτές τις δηλώσεις, όλα αυτά τα έντυπα. Μπορούμε να σας πούμε επίσης πόσο χρόνο αφιερώσαμε για κάθε επενδυτικό σχέδιο, συνολικά για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χωρίς να χρειάζεται έπειτα να διαιρέσουμε τη χρονική αυτή περίοδο ανά μέρα και χωρίς να χρειάζεται τελικά να κάνουμε μία κατάτμιση των δαπανών όσον αφορά τις κοινωνικές εισφορές ή όσον αφορά τους φόρους που καταβάλαμε. Δεν είναι ρεαλιστική η προσέγγιση αυτή όσον αφορά τις επενδύσεις τώρα. Προσπαθούμε να συγκρίνουμε πόσο στοιχίζει ένα χιλιόμετρο ποδηλατόδρομου από τη μία χώρα στην άλλη θα σας προκαλέσει εντύπωση το αποτέλεσμα, γιατί η το πιο ακριβό κόστος δεν είναι αναγκαστικά στις πιο ακριβές χώρες. Αν δούμε όμως την ε, μονάδα δαπάνης, τότε πραγματικά συντοποιούμε ότι ε, η τιμή πολλές φορές μπορεί να μην ήταν τόσο ραλιστική. ότι μπορεί να μην έγινε απαραίτητη έλεγχη, ότι μπορεί τελικά ο διαγωνισμός να δόθηκε σε έναν ανάδοχο ο οποίος δεν είχε να προτείνει την καλύτερη δυνατή λύση. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αυτού του είδους την τυποποίηση θα πρέπει να κάνουμε και να μην αναλωνόμαστε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες πώς ήταν ε, οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, πόσες μέρες διήρκησε η περίοδος ε, υποβολής προσφορών και το καθεξής. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα τελικά θα πρέπει να μετρούν περισσότερο και κυρίως πόσο, πόση κοινοτική χρηματοδότηση χρησιμοποιήθηκε η συγκεκριμένη επένδυση. Μήπως δεν θέλει και ο κύριος Κοράτσα να πει τίποτα. Παρακαλώ. τι περιλαμβάνει ο προπολογισμό του κόσμου. Μάλλον τι ύψος πρέπει να έχει, φυσικά. Θα έπρεπε να είναι υψηλότερος, αλλά αυτές οι αποφάσεις ε, ελήφθησαν τώρα στα πλαίσια των αποφάσεων για, το πολιετές, ε, για τις πολιετής δημοσιονομικές ε, προοπτικές. Τώρα βέβαια γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά η Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητα συγχωνεύτηκε με την Γενική Διεύθυνση Αγορών. Άρα αυτό σημαίνει πως υφίσταται καθοδικές πιέσεις ο προϋπολογισμός. Αλλά ο κόσμος είναι προϋπολογισμός συντονισμού που πρέπει να έχει αποτέλεσμα μόχλευση σε άλλους προϋπολογισμούς. Έτσι πρέπει να τον δούμε. Έτσι λοιπόν με την Next Tour προσπαθούμε να συζητήσουμε με αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις στις περιφέρειες που αποφασίζουν για τις διαρθρωτικές χρηματοδοτήσεις που εκεί τα ποσά είναι πολύ πιο υψηλά και στη συνεργασία με την Μάρε και τη Ρέτζιο προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και με τις γενικές διευθύνσεις Άγρι και Έμπλε είπα ότι οι 800 μας χιλιάδες ε, βοηθούν να δαπανηθούν τα 4 εκατομμύρια του έρασμος ΣΥΝ. Θα μπορούσα να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Εάν στο μέλλον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θελήσουν να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση του τουρισμού, φυσικά θα το επικροτήσω. Αλλά τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα αυτά που έχουμε. Συμφωνώ με την Ιζαμπέλα Ντελμόντε ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια, σαφήνεια, για τις επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίες, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κόσμο, ακόμη και οι μικρές. Γιατί το κόσμο χρηματοδοτεί συνεργασίες μικρομεσαίων. Για παράδειγμα, αν υπάρξει μία συνάντηση στην Κίνα τότε κάποιος φορέας, ε, κάποια συνεργασία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ε, θα μπορέσει να πάει στην Κίνα και να μιλήσει με τα ταξιδιωτικά πρακτορία των Κινέζων. Ακόμη και, για μια, ακόμη και αν για μια μικρή επιχείρηση φαίνεται τραβηγμένο, μπορεί να γίνει. Και όντως είναι και περίπλοκες οι διαδικασίες μας. Χρειάζεται απλούστευση πρέπει να είναι πολιτική προτεραιότητα της Επιτροπής. Και ο Επίτροπος Τίμερμαν εργάζεται επ' αυτού. Θέλει καλύτερες κανονιστικές διατάξεις. Ε, αυτό τον έλεγχο καταλληλότητας, το fitness check. Και για το site ε, έχει δίκιο η Σαμπέλα. Δεν είναι πάντα φιλικό προς τον χρήστη, αλλά έχουμε πολλούς περιορισμούς γιατί η Γενική Διεύθυνση κόμμα αποφασίζει για την δομή των ε, site μας ε, και μας δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δεν είναι εύκολο να είναι τόσο ε, εύκολη η χρήση του site λόγω των περιορισμών που μας θέτει η DGCOM. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ότι έληξε συζήτηση για την ειδική ομάδα τουρισμού. Παρακαλώ, η κυρία Γιάλα Σέντερ. Θαυμάσιες οι παρουσιάσεις. Αλλά με εξέπληξε το σχόλιο της κυρίας Μάισνερ. Γιατί επανέλαβε αυτό που πάντα ακούμε για τον τουρισμό. Αφού όλα πάνε καλά, γιατί να λάβουν ε, επιδοτήσεις. Ε, τότε να μην υπάρχει ε, λόγος μέσω του Horizon 2020 να χρηματοδοτήσουμε την ε, Bayer ή την ε, Ross. Το θέμα δεν είναι αν πάνε καλά τα πράγματα. Απλώς. Ο τουρισμός πάει καλά επειδή έχουν γίνει άλλα πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι πρέπει να παίζουν το βασικό ρόλο. Πρέπει να υπάρχει σωστός προπολογισμό πληρώνουμε πολύ περισσότερα για πολύ λιγότερο σημαντικού τομεί. Θα ήθελα λοιπόν να μην υπάρξουν αυτές οι προκαταλήψεις οι οποίες είναι παλιές. Θυμάμαι τον κύριο Φερχόγγεν που μου έλεγε στην Ολομέλεια «Κυρία Γιάλα, ούτε φράγκο για τον τουρισμό». Γιατί πάει μια χαρά. Ναι, έτσι νομίζουν ορισμένοι. Αλλά, ε, πρόεδρος, πρόεδρος. Εντάξει, κοιτάξτε, η μπλε κάρτα είναι 30 δευτερόλεπτα. Τώρα να μας πει η Γκεζίνε τι θέλει να πει, πώς να απαντήσει. Λοιπόν, όχι, δεν εννοούσα ότι δεν πρέπει να δοθούν περισσότερα για τον τουρισμό. Το είπα. Γιατί γενικά ορισμένες φορές ε, κάποια εγχειρήματα είναι τόσο επιτυχημένα που δεν χρειάζονται βοήθεια. Αλλά φυσικά συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μειώσουμε τις χρηματοδοτήσεις του τουρισμού. Αυτό ήθελα απλώς να πω. Πρόεδρος. Ωραία. Όλοι συμφωνούμε. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πολύ για την συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ για την απάντηση. Ευχαριστώ τους ομιλητές μας ε, για την παρουσία τους και για τις απαντήσεις την ερωτήση. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη. Ευχαριστώ και όλους τους παρευρισκόμενους που ήταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση για να ξανάρθουμε και να συνεχίσουμε την τόσο επιτυχημένη εργασία μας. Δεν έχω τίποτα για τα διάφορα τις ευχές μου προς όλους. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος 9 η ώρα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευχαριστώ πολύ. Τις καλύτερες ευχές μου.